Καλημέρα. όπω ξέρετε, ο κύριος Σικέσκι απουσιάζει. τουλάχιστον στην αρχή της συνεδρίασής μας και θα έρθει αν τα καταφέρει προς το τέλος της συνεδρίασης. Θα αναλάβω λοιπόν εγώ να προεδρέσω στην Επιτροπή Γεωργία σήμερα. Όπως αποφασίσαμε χθε και όπως γνωρίζετε, προτείνεται μια τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη για τις εκθέσεις που θα συζητήσουμε και θα ξεκινήσουμε από την έκθεση υπαριθμών 8, στη συνέχεια την έκθεση 9 και μετά το σημείο 7 και θα επανέλθουμε με την συνέχεια της ημερήσιας διάταξης με το 10 και το ε, σημείο 10 και 11. Λοιπόν, Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη μας έκθεση, το σημείο υπαριθμών 8, καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών στην αλυσίδα στην αγροτροφημική αλυσίδα μεταξύ επιχειρήσεων. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για το θέμα αυτό και όπως ξέρετε είναι μια έκθεση για την οποία ήδη έχει γίνει ανταλλαγή απόψεων και είχε έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Είχαμε όμως πολλούς συναδέλφους που ήθελαν το λόγο και δεν είχαμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε την ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Επομένως τώρα θα συνεχίσουμε για να μπορέσουν όλοι να εκφραστούν για την έκθεση αυτή. Σας προτείνω λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μπιουγή και την ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπιουγή που ε, είναι σήμερα μαζί μας. θα μας θέσει και πάλι το πλαίσιο ε, ε, μέσα στο οποίο κινείται αυτή η έκθεση. Μετά θα γίνει η συζήτηση με τους κυρίους και κυρίες βουλευτές και θα σας ξαναδώσουμε το λόγο για να κλείσετε το θέμα αυτό, κυρία Μπιουγή, εκ μέρους της Επιτροπής. Σας δίνω το λόγο, λοιπόν, για να ξεκινήσετε. Η κυρία Μπιουγή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή χαίρεται που ε, παρήσατε σήμερα εδώ για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν από μια εβδομάδα περίπου. Καταρχήν θα ήθελα να πω, την προηγούμενη φορά σημειώσαμε βέβαια πολύ προσεκτικά όλες τις ανησυχίες των Ευρωβουλευτών στην Επιτροπή σας. Ε, και έχουμε κατανόηση για τις ανησυχίες και ιδιαίτερα έχουμε κατανόηση για τα σημεία τα οποία τονίσατε για την επίπτωση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τονίστηκε αυτό το σημείο από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή μας εξάλλου. Καταρχήν Πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι θέλει να αντιμετωπίσει τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και ο υποψήφιος επίτροπος κύριος Χόγκαν, τον οποίο ε, είδατε στην ακρόαση στην Επιτροπή σας ε, και ο κ. Μπιακόφσκα ε, που μίλησε στην Επιτροπή Ήτρε και και οι δύο επίτροποι, ε, οι προτινόμενοι επίτροποι, ε, έχουν σαφή θέση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά τα σχόλια που έγιναν την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση από το 2010. Κάποιοι βουλευτέ είπαν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχει αλλάξει όμω η κατάσταση από το 2010. Έχει βελτιωθεί βελτιωθεί κάπως ε, η κατάσταση. Αναγνωρίζονται τα προβλήματα από όλους τους εμπλεκομένους. Ε, είναι γνωστό ότι υπάρχουν τέτοιες αθέμητες πρακτικές και τώρα το ποιες πρακτικές πρέπει ε, να καταπολεμηθούν είναι αυτό που συζητάμε. Υπάρχει επίσης η πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού και το ερώτημα είναι αν είναι επαρκής αυτή η πρωτοβουλία, αν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Η προσέγγιση της Επιτροπής είναι ότι υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία για την ε, εφοδιαστική αλυσίδα, διότι ξέρουμε ότι μπορούμε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Καταρχήν διαπιστώνουμε το πρόβλημα, οι εμπλεκόμενοι το αναγνωρίζουν και αποφασίζουν να καταπολεμήσουν τα προβλήματα, άρα αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά η ανακοίνωση λέει ότι δεν θα σταθούμε μόνο στην πρωτοβουλία αυτή για την εφοδιαστική αλυσίδα και πολλοί ευρωβουλευτέ δήλωσαν σαφώ ε, στην συζήτηση την περασμένη φορά ότι πρέπει να δούμε και τι άλλο χρειάζεται πέραν τη πρωτοβουλία αυτή για να αλλάξει η κατάσταση από τη, ε, από τη βάση. Η ανακοίνωση της επιτροπή εξετάζει και το θέμα του τι κάνουν τα κράτη-μέλη για την λήψη μέτρων. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη αν έχουν ανεξάρτητους φορείς που έχουν κάποια ε, εποπτεία των όσων συμβαίνουν επί τόπου. Τονίσαμε ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις καταγγελίες να γίνονται έρευνες από ανεξάρτητα, ανεξάρτητους φορείς και να ε, επιβάλλονται και αποτελεσματικές κυρώσεις. Μαρή Μαγκίνες έκανε την προηγούμενη φορά την ερώτηση πώς αξιολογεί η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα αυτών που κάνουν τα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω ότι αρκεί να κάνουμε καταμέτρηση των καταγγελιών. Αυτό δεν θα αλλάξει την κατάσταση. Αυτό που εξετάζει η Επιτροπή είναι τι συμβαίνει στην πράξη. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε να υπάρχουν λιγότερες αθέμητες πρακτικές, στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη είναι αποτελεσματικά και αποτρεπτικά. Ξέρουμε ότι η διαπραγματευτική δύναμη δεν είναι παντού ε, ισοδύναμη και δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικές οι κυρώσεις. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι η Επιτροπή δεν έχει πει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία νομοθετική ρύθμιση. Είπαμε ότι προς το παρόν δεν το βλέπουμε σκόπιμο και είπαμε ότι βραχυπρόθεσμα πρέπει να εξετάσουμε την πρωτοβουλία για την φοδιαστική αλυσίδα, να εξετάσουμε με αυστηρότητα το κατά πόσο λαμβάνουν μέτρα για την εφαρμογή τα κράτη-μέλη και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε περισσότερο μακροπρόθεσμα. Παραμένει ε, προτεραιότητα για την Επιτροπή το θέμα αυτό και όπως λέμε και στην ανακοίνωση αναλαμβάνουμε τη δέσμευση μέχρι το τέλος του 2015 να επανέλθουμε στο Κοινοβούλιο και να υποβάλουμε μια έκθεση για την πρωτοβουλία εφοδιαστικής αλυσίδας, τι έχει γίνει και πόσο αποτελεσματικές είναι οι κυρώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπουρή. Προτείνω τώρα να ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση. Η κυρία Μιούλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το πώς ε, η Επιτροπή αξιολογεί ε, το γερμανικό καρτέλ. Αυτό θα ήθελα εγώ κυρίως να ρωτήσω και αν υπάρχει κάποια γενικότερη εικόνα για το τι κάνουν τα κράτη-μέλη και πώς αντιμετωπίζουν τις εθνικές πρακτικές, πώς αξιολογούνται οι εθνικές πρακτικές και πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τη θέση των κρατών μελών. Τίθεται το θέμα του αν αρκούν αυτά τα οποία γίνονται ως εδώ θα πρέπει να λάβουν τα σωστά συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής ε, τα κράτη-μέλη κατά τον καρτέλ. Ευχαριστώ. Merci, Muller, monsieur. Σας ευχαριστώ κύριος Ούτεμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση. Νομίζω ότι μόνο 127 επιχειρήσεις έχουν ε, υποβάλει για την πρωτοβουλία αλυσίδας εφοδιασμού. Η Κομισιούν μπορεί να μου πει αν αυτό είναι επαρκές για να λειτουργήσει και τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να αυξήσει τον αριθμό αυτών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μποβέ έχει το λόγο. Πρόεδρε, άλλη μία φορά έρχεται η Κομισιόν εδώ με ένα κείμενο που δεν σημαίνει τίποτα άλλο, είναι απλώς ένα ευχολόγιο. Εφόσον δεν έχουμε νομοθετικό κείμενο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και σημειώνεται σωστά ότι στο πλαίσιο των συναντήσεων που έλαβαν χώρα διάφοροι φορείς δεν συμμετείχαν γιατί φοβήθηκαν τις συνέπειες. Ιδιαίτερα στον τομέα του κρέατος. έχουμε και το μυστικό της ε, καταγγελίας τέτοιων αθέμητων πρακτικών, το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται νομικά αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσουμε. Αν δεν έχουμε νομικό πλαίσιο δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Μόνο οι συζητήσεις δεν μας οδηγούν κάπου. Έχουμε πάντα μεγάλες συγκεντρώσεις. Σε προηγούμενη συνάντηση μιλούσαμε για συγκεκριμένες συνομαδοποιήσεις ε, ε, διανομέων Σήμερα πού βρισκόμαστε. Ποια είναι η απάντηση της Κομισιόν απέναντι στις πρακτικές αυτές. Χρειαζόμαστε αυτές και συγκεκριμένες απαντήσεις. Και άλλος ένας τομέας ο οποίος θα έπρεπε να εξεταστεί και δεν εξετάζεται είναι ο ρόλος των εξαγωγών των γεωργικών ο συνδυασμός με τα ενεργειακά διότι ο ανεφοδιασμός των εκμεταλλεύσεων είναι εξίσου σημαντικός με την αλυσίδα των τροφίμων. Και είχαμε επιμείνει στο Κοινοβουλίο και μάλιστα στο ψήφισμα με μεγάλη πλειοψηφία ακριβώς το θέμα του ανεφοδιασμού. Εδώ πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα, γιατί το κόστος της παραγωγής αυξάνεται, δεν υπάρχει διαφάνεια για τους παραγωγούς, οι οποίοι υποχρεούνται να προσαρμόζονται τα συστήματα των διανομέων. Πρέπει να πάμε πιο μακριά λοιπόν και η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι θα πάμε προς μια νομοθετική δεσμευτική πρόταση. Μάλιστα κύριε Μποβέ, ευχαριστώ. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και 24 χρόνια Είμαι μέλος και στο Γερμανικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 24 χρόνια που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα τα ίδια συζητάμε, την συγκέντρωση του εμπορίου. Και πολλές φορές έχω εκφράσει κριτική κατά του γερμανικού καρτέλ χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Δεν με εντυπωσιάζει λοιπόν που και πάλι ασχολείται ο τύπος και η συνάδελφος Μιούλερ το ανέφερε και στην Süddeutsche Zeitung ένα άρθρο στις 24 ε, Σεπτεμβρίου έλεγε ότι το καρτέλ ε, είναι ισχυρό, είναι μεγάλο και επιβάλλει τις τιμές του. Και ε, τα σούπερ έχουν πολύ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προχωρεί σε τέτοιο βαθμό αυτή η κατάσταση που απαιτούν από τους παραγωγούς των προϊόντων ε, ε, να κάνουν εκπτώσεις, να δώσουν μπόνους, ε, να προσφέρουν κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο θα προέβλεπαν οι συμβάσεις του και ως μέσο πίεσης χρησιμοποιούν ακόμη και απειλές ότι θα βγάλουν ε, τα προϊόντα των παραγωγών από τα ράφια των σούπερ μάρκετ και υπαγορεύουν τους όρους τους στους παραγωγούς. Ε, χαίρομαι που δημοσιεύονται τα άρθρα αυτά στον τύπο. Η Επιτροπή όμως τι κάνει, αφού η κατάσταση είναι γνωστή. Εδώ και δέκα χρόνια μόνο υποσχέσεις ακούω από την Επιτροπή. Oui, merci. ευχαριστώ. Η κυρία η κυρία Σέντρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ στα πορτογαλικά. Όχι, στα ισπανικά μιλάει η μιλητρία. Δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να μιλούμε για κωδίκους, ε, για κώδικες, με συγχωρείτε, πρακτικών εθελοντικούς. Πρέπει να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο δεσμευτικό. Από την άλλη, λείπει από τη συζήτησή μας το στοιχείο των μηχανισμών ώστε να είναι η επαγγελματική δραστηριότητα των παραγωγών, των γεωργών προσοδοφόρος, επαρκής για να επιβιώσουν δηλαδή. Διότι πάντοτε θα έχουμε τα φαινόμενα των πρακτικών αυτών από τις μεγάλες αλυσίδες στα τρόφιμα. Σας ευχαριστώ. Μιλάμε για τις αθέμητες πρακτικές των λιανικών εμπόρων σε σχέση με τους προμηθευτές και να ζητούμε λύσεις στο ενωσιακό επίπεδο. Σε οποιοδήποτε κράτος μέλος όπου υπάρχει διαφθορά και υπάρχει σε πολλές, είναι... προσπαθούν οι μεγάλοι λιανέμποροι να εξαγοράσουν τον επιθεωρητή, τον δημοπράτη και μπορείτε να έχετε ό,τι κανόνες και κανονισμούς θέλετε, αλλά αυτά τελικά δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα στην πρακτική. Στο Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό και ελπίζω ότι οποιαδήποτε νομοθεσία ενωσιακή θα ε, διασταυρωθεί με τη δικιά μας νομοθεσία. Έχουμε δημιουργήσει τη θέση του Δημοπράτη, έχουμε την κυρία ε, σαν εισαγγελέα τρόπον την σε αυτή την περίπτωση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη αλλά ο ρόλος της είναι να αποτρέψει τους λιανεμπόρους από ορισμένα από τα κόλπα τους. Αλλά θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δίωξης και να δείξει ότι έχει δόντια για να μπορέσουν οι λιανέμποροι κάπως να φοβηθούν. Έχουμε κάτι που το αποκαλούμε Επιτροπή Ανταγωνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιστεύω ότι η εντολή, οι εξουσίες πρέπει να μεταβληθούν διότι αποτρέπει τους προμηθευτές να συνενωθούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πραγματικά τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει ανισορροπία. Τα σούπερ μάρκετ επιτρέπεται να είναι ισχυρότερα μέσω των συνεταιρισμών και επιτρέπεται η ανισορροπία μέσω του νόμου τελικά είναι σαν να έχετε μία ποδοσφαιρική ομάδα με έξι παίκτες και μία άλλη με έντεκα. Εάν λοιπόν η Κομισιό είναι σοβαρή ε, και δύο υποψήφοι έχουν αναφορθεί, ε, υποψήφοι επίτροποι έχουν αναφερθεί, θα, θα πρέπει να προχωρήσουν με στένος. Αναρωτιέμαι όμως αν η Κομισιό είναι διατεθειμένη να το κάνει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κυρία Κόστιγκερ. Ευχαριστώ. Ήδη μου έκανε μεγάλη εντύπωση που στην παρουσίασή της η Επιτροπή είπε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση και αναφέρθηκε ως πρώτο σημείο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη προβλήματος, ε, ότι υπάρχει δηλαδή ε, υπάρχουν αθέμητες ε, πρακτικές. Με τέτοιες δηλώσεις όμως δεν βοηθάμε τους παραγωγούς που βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης πίεσης. Ε, οι αγρότες, οι παραγωγοί βρίσκονται υπό τεράστια πίεση και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα. Και την προηγούμενη φορά ε, είχα αναφέρει ότι οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ ε, πουλάνε το γάλα πιο φτηνά και από το νερό. Υπάρχουν πιέσεις οι οποίες είναι πραγματικά αφόρητες και απαράδεκτες θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε παραγωγούς, παραγωγούς λαχανικών ενδεχομένως, οποροκυπευτικών, όπου έχουν επιδεινωθεί ε, οι συνθήκες, ε, να, να δώσουμε τη δυνατότητα ε, τουλάχιστον να μπορούν να εκφράσουν τις καταγγελίες τους και να μην υφίστανται εκβιασμούς. και πρέπει τελικά να αντιμετωπίσουμε με ενεργό τρόπο το πρόβλημα. Φτάνει τελικά, ε, φτάνουμε στην κατάσταση η παραγωγή να αμείβονται σε επίπεδο χαμηλότερο του κόστους παραγωγής. Είναι πολύ σημαντικός τομέας και πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχουμε κάποια βελτίωση. Γι' αυτό λοιπόν Θέλουμε να δούμε τι δυνατότητες βελτίωσης έχει να μας προτείνει η Επιτροπή και για τα θέματα διαφάνειας. Ε, ευχαριστώ κυρία Κωστιγκερόν. Κυρία Μαγκίνες τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την περιγραφή των όσων συμβαίνουν και για την ανταπόκριση στο ερώτημα το οποίο έθεσα. Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι πέρσι το Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα κείμενο που ζήτησε μια αναθεώρηση της εθελοντικής πρωτοβουλίας μετά από ένα έτος εφαρμογής θέση σε ισχύ και ανεγνώρισε τα προβλήματα και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές λόγω των αθέμητων πρακτικών. Είναι ένα θέμα που έχουμε έντονη άποψη. Θέλω να θέσω δύο θέματα. Έχουμε την υπόθεση Τέσκο στον Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα. Τα κέρδη τους χειραγωγήθηκαν κρατώντας χρήματα τα οποία οφείλονταν στους προμηθευτές. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και νομίζω ότι πρέπει η Κομισιόν να το εξετάσει. Δεύτερον, πόσο σοβαρά ασχολείται η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Το δίκαιο του ανταγωνισμού ουσιαστικά καταστρατηγεί τις προσπάθειες αυτής της ε, Επιτροπής, διότι ενδιαφέρεται μόνο για τη χαμηλότερη τιμή. Και αυτό δεν είναι μια άποψη που υποστηρίζει την βιωσιμότητα της αλυσίδας τροφοδοσίας. Πόσο στενά συνεργάζεται λοιπόν η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τα θέματα που μας, ενδιαφέρονται, μας ενδιαφέρουν όσον αφορά τις αθέμητες πρακτικές. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και τον διαιτητή, ε, είναι σωστό να υπάρχει ένας διαιτητής ε, όσον αφορά την αλυσίδα τροφοδοσίας. Ε, τι νομίζει η Κομισιόν σε σχέση με το γεγονός ότι οι γεωργοί δεν έχουν υπογράψει τον κώδικα διοντολογίας διότι πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετά ισχυρός και δεν αντιμετωπίζει το θέμα του φόβου στην λυσίδα τροφοδοσίας που είναι έντονο. Νομίζω ότι η Επιτροπή πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο με αυτό το θέμα. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να είναι στην ατζέντα μας κάθε μήνα. Να ζητάμε ενημέρωση, τακτικότητα και να μην το ξεχνάμε είναι όσο σημαντικό όσο η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ επηρεάζει τη γεωργία, επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών που υποβαθμίζονται με αυτές τις πρακτικές. Παρακαλώ λοιπόν η Επιτροπή να ασχοληθεί σοβαρά μέλλοντικά. Ευχαριστώ. Σύμφωνο απόλυτα με την άποψή σας. Θα επανέλθω αργότερα. Ο κύριος Ρέμπεγκα εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Χαίρομαι που η Κομισιόν σημείωσε τις ανησυχίες μας σχετικά με τις αθέμητες αυτές τις Νομίζω όμως ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτήν την κατακαιρματισμένη προσέγγιση. Τα σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες αλυσίδες δρούν με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί να μην έχουμε μια οδηγία, λέει ο μιλητής, για να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ των παραγωγών και των διανομέων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βουαζού. Oui, Σας ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε η Γαλλία έχει ήδη πρόβλεψη νομοθετική για την καταπολέμηση των αθεμήτων πρακτικών. Μήπως υπάρχει κίνδυνος χαμηλότερο επίπεδο προστασίας για τη χώρα μας μέσω νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας ευρωπαϊκής. Η κυρία Ντελαή. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Μαγκίνες ε, και την κυρία Κιώστιγκερ γιατί και εγώ επιβεβαιώνω ως επαγγελματίας ε, ότι υπάρχει έντονη δυσκολία για τους παραγωγούς απέναντι στη διαδικασία. Είχα συναντηθεί με μια ένωση παραγωγών λαχανικών από τη Γαλλία σχετικά με μια αγωγή κατά αλυσίδας. Εννέα χρόνια η αγωγή αυτή κράτησε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτήν την ένωση των παραγωγών συλλογική αγωγή και όχι ατομική είναι σαφές ότι πρέπει να κινηθούμε ταχύτατα πλέον. Ακούσαμε ότι 24 χρόνια, πολλά χρόνια ακούμε αυτά τα ζητήματα. Εγώ ως ειδική στο χώρο τα παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και παρότι λέει ο κύριος Βουαζό ότι είναι επαρκές το νομοθετικό πλαίσιο, θα έλεγα εγώ ότι είναι ανεπαρκές. Γιατί πέραν των αποφάσεων των δικαστηρίων έχουν πάντοτε τη δυνατότητα οι αλυσίδε αυτέ να παρακάμψουν τι διατάξει και τον νόμο. Εγώ θα έλεγα να προσέξουμε ιδιαίτερα το ζήτημα αυτό που είναι ζωτική σημασία για του παραγωγού και την επιβίωσή του. νομίζω ότι από αυτού θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ επί του δικαίου του ανταγωνισμού γιατί στη Γαλλία πολύ πρόσφατα και εγώ ήμουν μαζί με αυτήν την ομάδα των παραγωγών που κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν ως για αθέμητες ε, διαδικασίες παραγωγής. Όταν λοιπόν έχουμε ενώσεις παραγωγών οι οποίοι τελικά πληρώνουν το ότι τολμούν να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν και να στραφούν κατά των, ε, των, ε, προσπα, αυτών προσπαθειών από πλευρά των διανομέων χάνουν έδαφος. Σας ευχαριστώ η κυρία Ριμπέρο έχει το λόγο. Eh, ευχαριστώ, καλημέρα σας. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να <clears throat> συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των μικρών αυτών φορέων χωρίς να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό. Συμφωνώ πολύ με την κυρία Μαγκίνηση η οποία λέει ότι η καταπολέμηση των αθέμητων αυτών πρακτικών πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Τώρα την προηγούμενη φορά εγώ είχα ήδη πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει κοινό νομοθετικό πλαίσιο. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτό. Ιδιαίτερα καθότι είμαστε και προχωρούμε όλο και περισσότερο σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και είναι πολύ ενδιαφέρον να κοιτούμε και ε, το πλαίσιο των ισχύων και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ακούσαμε και από συναδέλφους. <clears throat> Όπως ε, διαβάζουμε και στην ανακοίνωση, πολύ συχνά έχουμε προβλήματα ε, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως προς την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση αυτή και πρέπει να σκεφτούμε Αυτή την ιδέα του διαμεσολαβητή, του ombudsman, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, η Κοσμισιόν νομίζω ότι πρέπει να επανέλθει. Μάλιστα, σε ευχαριστώ κυρία Σχάιντα. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να παρέμβουμε πραγματικά, διότι όταν κοιτάμε τα κονδύλια τα οποία πηγαίνουν προς την αγορά και τις μεγάλες πολυεθνικές, αν συνεχιστεί η κατάσταση σε πέντε χρόνια, δεν θα υπάρχουν πια οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Και βεβαίως πρέπει να δούμε τι, τι είναι βιώσιμο, όπως τα φυτά, τα ζώα και ίσως πρέπει να κάνουμε έναν άλλο λογαριασμό διαφορετικό από τις πολυεθνικές που κρατούν τα χρήματα. Βλέπουμε ότι οι πολυεθνικές ουσιαστικά μέσω της νομοθεσίας κερδίζουν ακόμη παραπάνω χρήματα. Ε, και μια ισχυρή νομοθεσία στις κάτω χώρες στη χώρα μου ε, διέπει αν θέλετε τον ανταγωνισμό αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για την ε, παρουσίαση. Έχουμε ένα πρόβλημα ε, ουσίας εδώ πέρα. Έχουμε τα τραστ, την υπερσυγκέντρωση της διανομής. Υπό την γεωργική έννοια και υπό την έννοια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των γεωργικών. Το να προϋποθέτουμε ότι όλοι αυτοί έχουν καλές προθέσεις για να φτάσουμε σε εθελοντικές συμφωνίες είναι σαν να πιστεύουμε στους μάγους. Δεν μπορούμε όλα αυτά να το αφήσουμε στην καλή θέληση των ε, διαφόρων φορέων στην ε, τροφική αλυσίδα. Πρέπει να προχωρήσουμε κανόνε. Στην Ισπανία κάναμε. Προχωρήσαμε σε τέτοιο νομοθέτημα και το οποίο ορίζει πλαφόν για τις καταβολές στους ε, διανομές. Και είναι αυτό που ζητώ από την Κομισιόν. Μιλούμε για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Υποφέρει η μικρή και μεσαία επιχείρηση στον τομέα, πρέπει να το επιλύσουμε. Επίσης έχουμε αυτή την εσωτερική αγορά η οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να λειτουργεί και αυτή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριο Μισελ choses. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά τύχη εξετάζουμε δύο πράγματα που είναι πολύ συμπληρωματικά. Αφενός τις ε, αθέμητες πρακτικές ε, και το θέμα γενικώ ε, της ανταγωνιστικότητας της κοινή γεωργικής πολιτικής. Τώρα έχουμε τη λειτουργία της διατροφικής αλυσίδας, των μεγάλων διανομέων, των μεγάλων αλυσίδων στην συμπίεση του συστήματος. μειώθηκε 16% η τιμή των, ε, των, ε, Dans une guerre commerciale. των ζυμαρικών. Δηλαδή οι μεγάλες αλυσίδες είναι έτοιμες να κάνουν τα πάντα για να κατεβάσουν την τιμή. για να κερδίζουν σε ανταγωνιστικότητα έναντι των άλλων επιχειρήσεων τι οποίε ανταγωνίζονται. Και οι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσεις ποιοι είναι, είναι τελικά το θύμα του συστήματος αυτού. Και ποιο θα εκμεταλλευτεί την πιθανή χρεοκοπία τους. άλλε ακόμα πολυεθνικές εταιρείε, οι οποίε θα παρέμβουν, θα μπουν στην αγορά και θα καταστρέψουν ακόμα περισσότερε θέσει απασχόληση. Είμαστε εκεί να προστατεύσουμε του ε, καταναλωτέ αλλά και τι θέσει απασχόληση. οι επιχειρήσει οι γεωργικέ έχουν θέσει επανειλημμένο το πρόβλημα σχετικά με θέσεις απασχόλησης χαμηλή ε, ειδίκευση, αλλά πολύ σημαντικέ υπό την έννοια ενό ελάχιστου εισοδήματο, αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη στι συζητήσει μα, το θέμα δηλαδή τη απασχόληση και των συνεπειών αυτού του ανταγωνισμού χωρίς όρια και χωρίς κανόνες οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων είχαν αποφασίσει ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν πρέπει να παρακολουθεί από νέα νομοθετική πρωτοβουλία, από πρωτοβουλία καινούργια, καθότι δεν έχουμε πρόταση. Αλλά είναι μια ανταπόκριση της Κομισιόν στο αίτημα του Κοινοβουλίου. Έχω την εντύπωση αυτή η ανακοίνωση. Σας ευχαριστώ κύριε Νταντάν, κύριος Ρούπε. E, e, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα που αντιμετωπίζουμε. Και μάλιστα υπό το φως του ρωσικού εμπάργου διαπιστώνουμε ότι οι τιμές έχουν μειωθεί περισσότερο από 30% αλλά δεν έχει αλλάξει ε, η τιμολόγηση από αυτούς που κάνουν τη μεταποίηση ή στα σούπερ μάρκετ. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή. Ε, Παρ' όλα αυτά, οι μεταποιητές και οι λιανοπολιτές είναι αυτοί οι οποίοι καρπούνται την βοήθεια που εμείς δίνουμε στους παραγωγούς και τελικά απομένει πολύ μικρό μερίδιο στον παραγωγό. Μόλις που επιβιώνουν οι παραγωγοί. Και αν δεν υπάρξει νομοθεσία για να ρυθμίσουμε αυτές τις διαδικασίες θα συνεχίσουμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Ίσως αυτή η μελλοντική οδηγία που συζητάμε δεν μπορεί να είναι τέλεια από την αρχή και μπορεί να βελτιωθεί αργότερα. Πρέπει πάντως ε, να εμπλακούν και οι οργανώσεις των αγροτών στην προετοιμασία της οδηγίας αυτής. για να μην επωφελούνται οι μεταποιητές και οι λιανοπολιτές από τα μέτρα τα οποία εμείς λαμβάνουμε προς όφελος των παραγωγών. Στη Λιθουανία έχουμε παραδείγματα όπου δόθηκε μεν ενίσχυση σε αγρότες, αλλά τα χρήματα κατά βάση πήγαν στους πιο δυνατούς κρίκους της αλυσίδας τροφίμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νόιχλα. Η κυρία Όντως επικρατεί φόβος ε, μεταξύ των παραγωγών. Υπάρχει τεράστια πίεση. Ε, οι τιμές dumping ε, επιβάλλονται σε οικογένειες παραγωγών και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα, διότι μεγάλες εταιρείες, μεγάλοι όμιλοι, αν ένας παραγωγός δεν δράσει σύμφωνα με τις οδηγίες του, να τον αλλάξουν, να σταματήσουν να προμηθεύονται από αυτόν. Και όλο και περισσότερο συνεχίζεται αυτή η πρακτική. Θυμάμαι την την εποχή που υπήρχε κάποια απεργία στον τομέα του γάλακτος στη Γερμανία και δεν ε, γίνονταν παραδόσεις γάλακτος, άρχισαν να φέρουν γάλα από άλλες περιφέρειες. Υπάρχει και δυνατότητα ε, εναλλαγής προϊόντων ε, και η κατάσταση του dumping ε, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις οικογενειακές επιχειρήσεις διότι πιέζονται ε, από τις μεγάλες εταιρείες που τους λένε ότι θα αλλάξουν τον παραγωγό εάν δεν συμμορφωθούν με τους όρους τους. Merci. Ευχαριστώ. Η κυρία Έγαν. Sí, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η Κομισιόν αν θέλετε δεν με ικανοποίησε πραγματικά με την εξή έννοια. Δεν χρειάζεται μόνο να έχουμε συστάσεις για διάφορα προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει. Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο κανονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλιώς δεν θα υπάρξει ε, συγκεκριμένη λύση, δεν θα ξεπεράσουμε τις αθέμητες πρακτικές. Ε, παραγωγοί φοβούνται να ανακοινώσουν τις ε, καταχρήσεις, ο φόβος κυριαρχεί στους παραγωγούς, τα θύματα αυτά χάνουν τα χρήματά τους, δεν μπορούν να έχουν ρευστότητα, η Κομισιόν πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται. Είναι κρίμα ότι στο Συμβούλιο πριν από μερικούς μήνες δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν ε, βάσει των προτινόμενων ιδεών. Η Ισπανία έκανε συγκεκριμένες προτάσεις, το Συμβούλιο δεν ακολούθησε και ακούσαμε τον υποψήφιο επίτροπο την περασμένη εβδομάδα, μας είπε ότι ήταν διατεθειμένος να ακολουθήσει μια πρωτοβουλία και να νομοθετήσει. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι πιστεύουν οι υπηρεσίες της Κομισιόν σε σχέση με αυτό που είπε ο υποψήφιος επίτροπος. Ίσως είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να γίνει. Πρέπει να συμφωνήσουμε για μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Αναγκαστικό χαρακτήρα, ώστε να δώσουμε τον μηχανισμό στα κράτη-μέλη να υπερασπιστούν τους παραγωγούς. Πιστεύω ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να προσδιορίσει τις πρακτικές που πρέπει να υποστηρίξουμε και πρέπει ακόμη να επιβάλλει ελέγχους σε όλα τα κράτη-μέλη με πραγματικές κυρώσεις για αυτούς που καταχρώνται την θέση τους. Πιστεύω ότι η Κομισιόν πρέπει να ακολουθήσει αυτή την, αυτόν τον προσανατολισμό. Ο, ο, ο Επιτροπός μας το είπε την περασμένη εβδομάδα, θέλουμε πράξεις. Ευχαριστώ. Ο Πόλο Ντικάστρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου φαίνεται ότι η θέση της Επιτροπής μας είναι σαφής. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και το έγγραφο της Κομισιόν είναι πολύ αδύναμο. Ελέγχθησαν πολλά πράγματα σε σχέση με το επίπεδο συγκέντρωσης παραδείγματος χάρη. Όσον αφορά τους διανομής που είναι τελείως άνισο σε σχέση με τις μικρομεσαίες. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια νομοθεσία ευρωπαϊκή για να αποφύγουμε, να αποφύγουμε τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Και αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας θα πρέπει να εναρμονίσουμε αυτούς τους κανόνες. Αλλιώς η στρέβλωση του ανταγωνισμού θα συνεχίσει. Συμφωνώ με τον Μισελ Ντοντά. Χρειαζόμαστε έκθεση πρωτοβουλίας. Θέλουμε δέσμευση της Κομισιόν. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Επιτροπή Γεωργίας, αφορά και άλλες επιτροπές. Θέλουμε μία δέσμευση από τον Γιούγκερ για να ρυθμίσουμε το πρόβλημα. αλλιώ. θα συνεχίζουμε να λέμε και να κλεγόμαστε για τι αθέμητε πρακτικέ και τα κράτη-μέλη δεν θα κάνουν τίποτα. Ο uh, κύριος Μπάνιν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να προσθέσω και εγώ τη δική μου φωνή ζητώντας έναν ε, εθελοντικό κώδικα από την Κομισιόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι η σημασία της αντιμετώπισης του φαινομένου των ανθέμινων πρακτικών από κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ε, και χονδρικών πολιτών είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Είχαμε εμείς έναν κωδικό που εισήχθη από την κυβέρνηση Labour το 2010, το οποίο παρέχει στους συνεταιρισμού και τους αγρότες ε, με κάποιο είδους δυνατότητα καταγγελίας. Το οποίο αποτρέπει αντιμέτρα από πλευρά των αλυσίδων όταν έχει υποβληθεί μια τέτοια καταγγελία. Και υπάρχει αυτή η προστασία για τους Βρετανούς γεωργούς, αλλά δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένως θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση υποβολής μιας ε, καταγγελίας και μετά μια ένα αντιμέτρο, δηλαδή να καταλήγει προς, το, προς εις του αυτή η καταγγελία που έχει υποβάλει τελικά κάποιος ε, παραγωγός ή κάποια ένωση παραγωγών. Και αυτό που συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι καθίστε προφανές είναι ότι υπάρχει μια καλή πρόθεση. Προσπαθούμε να έχουμε ένα ισότιμο παιχνίδι για όλους εδώ. Αλλά έχουμε και αρνητικές συνέπειες καμιά φορά από αυτές τις προσεγγίσεις μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιό να προσέξει πολύ τι αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει αυτό που προτείνει. Δεν χρειάζεται να είναι ενιαίο το σύστημα για όλους το ίδιο. Δεν χρειάζεται όλοι να κάνουν αυτό που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ίσως να χρειάζεται μια πιο ευέλικτη light προσέγγιση αλλά για τη δημιουργία ενός ισότιμου παιχνιδιού είναι ένα σημαντικό βήμα αυτός ο κώδικας. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε από την Κομισιόν τι θα μπορούσε να κάνει για να αντιμετωπίσει τις αθέμητες αυτές πρακτικές ε, κάποιων αλυσίδων και σούπερ μάρκετ ενάντια των παραγωγών. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Όζριν. Äh, πρέπει να πω ότι με ενοχλεί που συνεχώς κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και η κατάσταση αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει. Υποστηρίζω την κυρία Μακίνες λοιπόν σε αυτά τα οποία είπε. Θα πρέπει να καταβάλουμε λίγο πιο εντατικές προσπάθειες και συμφωνώ και με τον Πάολο Ντεκάστρο. Θα πρέπει ε, να κάνουμε συζητήσεις που θα φτάσουν μέχρι τον κύριο Γιούγκερ γιατί θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν αρκεί να κάνουμε εκκλήσεις χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και πριν από δύο-τρία χρόνια είχαν γίνει συζητήσεις για το πακέτο των γαλακτοκομικών και αυτές έδειξαν ότι πουθενά δεν οδηγούσαν οι συζητήσεις Τελικά τι είπαμε, ότι δεν ε, πρέπει και να παραοργανώνονται οι παραγωγοί, γιατί υπάρχει και στρέβλες του ανταγωνισμού. Μία συζήτηση του παραλόγου. Όταν προσπαθούσαν ε, να οργανωθούν οι αγρότες για να ε, προωθήσουν τα προϊόντα τους, λέγαμε ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ δεν μπορούσαν να λαμβάνουν μέτρα για να προμηθεύονται από άλλους προμηθευτές. Υπάρχουν, υπάρχει μια αθέμητη συμμαχία κατά των παραγωγών πολλές φορές και πρέπει να δούμε τα συγκεκριμένα προβλήματα. τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις διατάξεις που προτείνονται και εγώ έχω την εντύπωση ότι ποτέ, πολλοί δεν τα θέλουν αυτά τα οποία προτείνουμε. Βλέπουμε ότι μειώνονται οι τιμές ε, και αν φτηνίνουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ ε, θα ανοίξει το πεδίο για κατανάλωση άλλων ειδών διατροφής παράλληλα με τα γεωργικά προϊόντα. Βελτιώνεται δηλαδή η κατάσταση για τον καταναλωτή. Οπότε τηρούμε σιγή για τα θέματα των αγροτών. Ευχαριστώ κύριε Ογλίν. Έχουμε ακόμη τρεις ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο και προτείνω να κλείσουμε τη συζήτηση μετά τους τρεις αυτούς ομιλητές και να ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία Περέη. Ο κύριος Γλέζος έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προβλήματα είναι πολλαπλά Ξεκινάω από το πρώτο πρόβλημα του αθέμητου ανταγωνισμού, της εμπορίας που αποσκοπεί στην κερδοσκοπία. Πώς εμείς θα καταργήσουμε την κερδοσκοπία των εμπόρων. Εδώ θέλω κάτι συγκεκριμένο από την πλευρά σας για να μην αρχίσω να λέω εγώ τη μια γνώμη και άλλο την άλλη. Γνώμη πώς θα καταργηθεί η κερδοσκοπία ως τώρα δεν υπάρχει. Δεύτερον, <coughs> είναι ο εκτοπισμός των μικρών γεωργών από μεγάλους ομίλους αγροτών από τα καρτέλ. Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα τρίτο πρόβλημα που αφορά τη γνησιότητα των τροφίμων των γεωργικών ειδών. Όταν νερώνω το κρασί νοθεύω. Όταν βάζω πέτρα στα φασόλια και στις φακές για να βαρύνουν περισσότερο κάνω μια μορφή νοθείας. Όταν κλωνοποιώ όχι τα ζώα μονάχα αλλά την κολοκυθιά για να παράγει καρπούζι κάνω νοθεία. Όταν όπως παραδείγματος χάρη γίνεται με τις τεράστιες ποσότητες μουστου από τη Σαντορίνη που μέσω την νησίας έρχονται στη Γαλλία και παρουσιάζονται ως κρασί μπορντό. Όταν πίνετε εσείς το κρασί μπορντό πίνετε μουστο από την Σαντορίνη και έχει μεγάλη αξία και ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων. Σε πολλά μέρη και στην πατρίδα μου την Ελλάδα χρησιμοποιούνται σκλάβοι για την παραγωγή τροφίμων. Για όλα αυτά τα θέματα ποια συγκεκριμένα μέτρα παίρνουμε. Θέλω συγκεκριμένη απάντηση σε αυτά. Merci. La parole à Monsieur Ευχαριστώ κύριε Ashworth. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ε, έχω πολλά περιστατικά θέμη των πρακτικών στον κλάδο και καταλαβαίνω πάρα πολύ τα προβλήματα που υπάρχουν από την πλευρά των παραγωγών και ιδιαίτερα των μικρών παραγωγών. Παρόλα αυτά, η συμβουλή μου προς την Επιτροπή θα ήταν να χρησιμοποιήσει νομοθετικές ρυθμίσεις μόνο ως τελευταίο μέτρο και το λέω διότι δεν μπορούμε να παραμερίσουμε τη δυνάμεις της αγοράς και τέτοιου είδους νομοθεσία πάντοτε θα είναι εύκολο να την παραβούν όσοι θέλουν να την παραβούν. Πρέπει να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τις βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας εφοδιασμού και έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα εθελοντικής ε, συμμόρφωσης που λειτουργούν πολύ σωστά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς να συνεργάζονται για να μην είναι απλώς παραγωγή ε, γεωργικών προϊόντων, αλλά να μπορούν να έχουν την κρίσιμη μάζα που θα τους οδηγήσει να έχουν προστιθέμενη αξία και θα τους οδηγήσει και σε μια κατάσταση ισορροπίας της αγοράς. Και κατά παρόμοιο τρόπο στην ε, λιανική πώληση θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις σωστές σχέσεις, να ε, δούμε ποιοι είναι η τοπική, περιφερειακή παραγωγή, να υπάρχει μια σχέση που θα οδηγήσει σε κοινέ επενδύσει και θα είναι ε, επιμεριζόμενοι και οι κίνδυνοι και επιμεριζόμενα και τα κέρδη. Τέτοιου είδου σχέσει πρέπει να έχουμε ε, και για τι σχέσει αυτέ θα πρέπει να υπάρχει και σωστή εποπτεία. Η εποπτεία θα πρέπει να γίνεται από ένα ανεξάρτητο διαμεσολαβητή, ένα ανεξάρτητο διαιτητή και θα πρέπει το ισχυρότερο όπλο αυτού του διαιτητή να είναι το ότι θα μπορέσει να καταγγείλει συγκεκριμένους παραβάτες. Αυτό είναι το ισχυρότερο όπλο και Νομίζω ότι ένας διαμεσολαβητής θα ήταν η καλύτερη πρακτική. Βέβαια, όταν υπάρχει απροθυμία συμμόρφωσης και από τις δύο πλευρές της τροφιμικής αλυσίδα, ίσως χρειαστούμε νομοθετικέ ρυθμίσεις, αλλά θα παρακαλέσω πολύ να το κάνουμε με μεγάλη φιδό. Ευχαριστώ. κυρία Πέτρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η μικρομεσαίοι παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να έχουν δυνατότητα σωστή τιμολόγηση των τροφίμων τους. Και έχω δύο ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Όταν υπάρχουν αθέμητες πρακτικές και βλέπουμε ότι κάποιοι γίνονται πλουσιότεροι ενώ άλλοι γίνονται φτωχότεροι, τι μπορεί να κάνει η κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να έχουμε ισότητα μεταξύ των παραγωγών και ισότητα μεταξύ παραγωγών και λιανικού εμπορίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές ε, που τοποθετήθηκαν. Το ζήτημα αυτό είναι προφανές ότι είναι πολύ σημαντικό των αθέμητων πρακτικών και εγώ προσωπικά πιστεύω πως πολλοί από εσάς παρότι που θα, πρέπει σε επόμενους μήνες να προετοιμάσουμε την επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αυτή η πτυχή είναι μια πτυχή επί της οποίας θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και εκεί η πρόταση της κυρίας ε, Μαγκίνες να υπάρξει τακτική παρακολούθηση μου φαίνεται πολύ χρήσιμη. Δεν ξέρω αν πρέπει να περάσουμε από μια πρόταση πρωτοβουλίας άκουσα και τα σχόλια του κυρίου Νταντά, πέρα από τα γεωργικά καθαρά προβλήματα, βλέπουμε ότι η πτυχή αυτή υπερβαίνει τα στενά προβλήματα της αγροτικής παραγωγής. Και πρέπει να δούμε τις πρακτικές αυτές και το αθέμητό τους, αλλά πρέπει να πάμε προς μία προσέγγιση νομοθετικής παρέμβασης ώστε να δίνουμε τα μέσα ελέγχου. Πρόκειται πάντως για ένα ουσιώδες ζήτημα και πρέπει να ασχοληθούμε στενά, να εξετάσουμε στενά το ζήτημα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, να δώσω το λόγο στην κυρία Μαγκίνης πρωτού επιστρέψω το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που επανέρχομαι. Έχω δύο συγκεκριμένες προτάσεις να υποβάλω σε σχέση με το τι θα κάνουμε μετά. Είναι η Επιτροπή ΙΝΚΟ και όχι η Επιτροπή Άγκρη που θα απαντήσει στην ανακοίνωση αυτή. Εγώ ζήτησα να έχουμε μία γνωμοδότηση, δεν ξέρω ποια είναι η θέση των συντονιστών, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και εμείς μία τοποθέτηση σε απάντηση αυτής της ανακοίνωσης της Κομισιόν. Επίσης, εγώ έγραψα στον κύριο Γιούνκερ ζητώντας του να θέσει το θέμα αυτό της τροφικής αλυσίδας υπό τη δικαιοδοσία της Επιτροπής Αγκρή. Έλαβα μία ασαφή και ασθενή απάντηση, είπε ότι θα το συζητήσει το θέμα με τον νέο Επίτροπο, αλλά ε, πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να γράψει ως Επιτροπή στον κύριο Γιούνκερ και να του ζητήσει να κάνει αυτό που είπα, ότι θα πρέπει να εμπίπτει στην εντολή της Επιτροπής Γεωργικών Ζητημάτων. Ναι, για να δούμε πρόεδρε αν μπορούμε να προχωρήσουμε τελικά με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε την πρότασή σας. θα ζητήσουμε από τον κύριο Φρέσκι να βάλει το θέμα αυτό στις επόμενες συνεδριάσεις των συντονιστών ώστε να πραγματοποιηθεί ουσιαστική εργασία. Κύριε Τζουρί, νομίζω ότι τα θέματα είναι σαφή. Μέσω των παρεμβάσεων είδατε πόσο ανησυχία υπάρχει και πόσο σπουδαίο είναι το ζήτημα. Συνεπώς, έχουμε όλοι ευθύνη. Γι' αυτό και σας δίνω το λόγο για να μας πείτε την απάντησή σας. Θα είμαι πολύ σύντομη. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τα μέλη για τα σχόλιά τους, τις παρατηρήσεις τους, τις ερωτήσεις τους. Βεβαίω η Κομισιόν αντιλαμβάνεται πόσο έντονα τοποθετήσετε ε, σε αυτό το θέμα. Θα το συζητήσω και με τους άλλους συναδέλφους στην Κομισιόν, αλλά όπως είπε η κυρία Μαγκίνες, πρέπει να μιλήσουμε και με άλλες επιτροπές για αυτό το θέμα, διότι τελικά, αν πρόκειται να υπάρξει νομοθεσία, πρέπει να είναι θέση ολόκληρου του Κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να έχετε περαιτέρω διάλογο με τα, τις άλλες επιτροπές. Ε, θα δώσω πέντε σύντομες απαντήσεις όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Η Φράου Μίλλερ αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησης στο γεγονός ότι το Bundeskartell στη Γερμανία είναι πολύ δραστήριο. Βλέπουμε επίσης και σε άλλα κράτη-μέλη τα συστήματα να ενισχύονται και αναφέρομαι ειδικότερα στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία που πολύ πρόσφατα μετέβαλε την νομοθεσία της. Η Φράου Μιούλερ ρωτήσατε αν η Κομισιόν αντιλαμβάνεται τόσα συμβαίνουν στα κράτη-μέλη. Ναι, το γνωρίζουμε, έχουμε εκδώσει μια νομική μελέτη ε, μαζί με την ανακοίνωση που σας δίνει μια σύνοψη της κατάστασης και βεβαίως ευχαρίστω να σας ε, ενημερώνουμε με κάθε εξέλιξη αλλά σας παρακαλώ διαβάστε τη νομική μας μελέτη δεύτερον το Δεκέμβριο θα έχουμε μια συνάντηση όλων ε, των αρχών εφαρμογής του δικαίου ε, από τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της κυρίας Τάνκομ από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενθαρρύνουμε μια ανταλλαγή καλών πρακτικών και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια τουλάχιστον σε σχετικά με όσα συμβαίνουν στα κράτη. Όσον αφορά την αλυσίδα τροποδοσίας ε, ένας βουλευτής είπε ότι θέλουμε ένα κώδικο ε, εθελοντικό δεοντολογίας ε, στην Ευρώπη. Υφίσταται αυτό. Δεν προσπαθούμε να τους βάλουμε όλους σε ένα καλάθι. Δεν είναι ένα σύστημα και μία διαπίστωση. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ κρατομελών. Υπάρχει όμως κώδικας δεοντολογίας εθελοντικός στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας Ολλανδός βουλευτής ε, ρώτησε αν υπάρχουν πολλοί προσυπογράφοντες. Πολλοί λιανέμποροι έχουν υπογράψει, αλλά όχι αρκετοί. Ε, θα θέλαμε περισσότερες μικρομεσαίες και θα θέλαμε και η παραγωγή βεβαίως να υπογράψουν, να συμφωνήσουν δηλαδή. Πολλές φορές ελέγχθη ότι η νομοθεσία είναι ο μόνος τρόπος να λυθεί το πρόβλημα. Ορισμένα μέλη αναφέρθηκαν και σε προβλήματα που ξεπερνούν τις αθέμητε πρακτικές. Αντιλαμβάνεται η Κομισιόν ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες στον τομέα, Αναφερθήκατε και στα προβλήματα με τις ρωσικές κυρώσεις, την παρακράτηση πληρωμών. Μπορεί βεβαίω να έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα λόγω αθέμητων πρακτικών, αλλά πρέπει να εξατομικεύσουμε την προσέγγιση. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα διαμίας. Μιλάμε για τις αθέμητες πρακτικές. Βεβαίως αυτές οι αθέμητες πρακτικές ε, ρεάζουν πολύ αρνητικά ειδικά τις μικρομεσαίες και το έχουμε αυτό κατά νου βεβαίως. Τέταρτον, διάφορα μέλη είπαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε μόνο ένα κώδικα, χρειαζόμαστε αποτρεπτική πολιτική. Ακριβώς αυτό αναγνωρίζει η ανακοίνηση της Κομισιόν. Δηλαδή αυτοί οι κώδικες δεν φτάνουν για να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα. Υπήρξε επίσης το θέμα ε, του διαιτητού. Κάποια μέλη είπαν ε, να υπάρχει ομπουτσμαν ε, στο επίπεδο το εθνικό. Συμφωνούμε με αυτό, βλέπουμε πλέον εκτίματα. Αλλά κράτη-μέλη είπαν ε, ότι πρέπει να έχουμε έναν διαιτητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να σκοπίσουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι πολλές από αυτές τις υποθέσεις έχουν σχέση με τις περιστάσεις. Χρειάζεστε κάποιον επιτόπου που να μπορεί να αναλύσει και να ερευνήσει επιτόπου. Σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα η Κομισιόν δεν έχει αυτές τις εξουσίες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεχόμαστε ότι η κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια μέσω των αρχών εφαρμογής των κανόνων αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω πριν πάμε στην νομοθεσία. Μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με σχετική νομοθεσία, όπως είπαν ορισμένοι βουλευτές. Ε, ε, δεν είναι εύκολο η νομοθεσία να εφαρμοστεί σωστά ή να καλύψει τα πάντα που χρειαζόμαστε. Υπήρξαν και συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την συγκέντρωση και το ρόλο του, της υπηρεσίας ανταγωνισμού. Ε, οι συνάδελφοί μου είναι εδώ και θα σας μιλήσουν σήμερα για την ΚΑΠ. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα να σας απαντήσουν και πάνω σας τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ όλα τα μέλη. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες σας και θα επανέλθουμε για να σας ενημερώνουμε αν το επιθυμείτε. Ευχαριστώ. Oui, merci, Madame Je crois... θα επανέλθουμε και δεν έχει κλείσει το ζήτημα. Ας μην ξανέξουμε την συζήτηση. Ας μην προεκτείνουμε μάλλον τη συζήτηση. Απλώς θα, θα δώσω για μια τελευταία φορά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Και αυτή είναι και η απάντησή μου προς την Επιτροπή. Χρειαζόμαστε αυστηρούς κανόνες, του οποίους πρέπει να συζητήσουμε. Το είδαμε και τα θέματα της περιαγωγής. Αν δεν είχαμε λάβει αυστηρά μέτρα, θα συνέχιζαν να πληρώνουν πανάκριβα την περιαγωγή οι καταναλωτές. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυστηρούς κανόνες που να ισχύσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διαφορετικά δεν πρόκειται να επιτύχουν αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, ας κλείσουμε προς το παρόν αυτό το σημείο είναι μια πρώτη βεβαίω εξέταση απλώς του ζητήματος και ας περάσουμε στο δεύτερο σημείο τη διατάξεως που συνδέεται άμεσα. Θα ζητήσω από τον κύριο Πολ Σίζα από πλευράς τη Κομισιόν να μας παρουσιάσει τα θέματα του ανταγωνισμού ή στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. και δύο κυρίω σημεία. Οι κατευθυντήριε γραμμέ ε, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στο άρθρο 206 οι συνάδελφοι που έχουν συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση θα τοποθετηθούν επί την συζήτηση που έχει ήδη γίνει επί των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών της ε, ΚΟΑ για να είμαστε σίγουροι ότι εφαρμόζουμε αντίστοιχους κανόνες από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ώστε να μην έχουμε διακρίσεις. Το δεύτερο σημείο είναι μια μελέτη που θα υποβληθεί, που θα παρουσιαστεί μάλλον που έγινε στις 2 Οκτωβρίου και στην οποία δεν συμμετείχαμε διότι έγινε την ίδια στιγμή με την ακροματική διαδικασία για τον, κύριο, για τον υποψήφιο επίτροπο κύριο Λόγκαν. Αφορά αυτό πάντως στον αντίκτυπο του λιανικού εμπορίου και στις καινοτόμες στρατηγικές στον τομέα των ε, τροφίμων. Ο κύριος ε, Σίζαρ έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει αυτό το θέμα. Νομίζω 10 λεπτά πρέπει να σας φτάνουν για να ανοίξουμε μετά τη συζήτηση. Σχετικά με την εφαρμογή λοιπόν αυτών των βασικών κανόνων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Είναι με χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα για να σας παρουσιάσω αυτά τα δύο ζητήματα. Ίσως να θυμάστε ή να γνωρίζετε ότι τον Ιούλιο είχα αποστείλει μια επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής σας ε, σχετικά με το έργο της ε, ΓΔ ΚΟΜΠ ανταγωνισμού θεωρώντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την μελλοντική σας δουλειά. Με χαρά λοιπόν βρίσκομαι όπως έλεγα εδώ για και έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω αυτά τα ζητήματα. Τώρα για το σχέδιο των ε, κατευθυντηρίων γραμμών των εξαιρέσεων ε, κανόνων ανταγωνιστών για το ελαιόλαδο, ε, το κρέας και Um, as you know, in 2013, the cap reform... και τις αεροτρές καλλιέργειες. Όπως ε, γνωρίζετε έχουν επέλθει διάφοροι τροποποίησεις του κανονισμού της ΚΑΠ σχετικά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε τομέα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αλλά μένοντας σε μια προσέγγιση της αγοράς market-based approach. Τώρα έχουμε τη νέα εξαίρεση για τις κοινέ πωλήσει από πλευρά παραγωγών να υπογραμμίσω τις βασικές αλλαγές. Οι νομοθέτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς αντιμετώπισαν εδώ και πολύ καιρό δύο ζητήματα. Πώς μπορούν οι καλλιεργητές να έχουν περισσότερα από την αγορά όταν έχουν λιγότερα ως δημόσια ενίσχυση και καθότι έχουν πολύ μικρή διαπραγματευτική ικανότητα και αντιμετωπίζουν τεράστιο ανταγωνισμό. Και όπως είπε ένα μέλος της Επιτροπής σας πριν από λίγα λεπτά, η λύση που προβλέπουμε θα έχει κάποια δόντια, θα έχει κάποια ισχύ δηλαδή. Τώρα η συμμόρφωση προς την εξαίρεση βασίζεται στους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής στο άρθρο 39 της ειδικής και όχι στο 101 των γενικών διατάξεων ανταγωνισμού. Υπό την έννοια αυτή λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ε, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε τομέα και κάθε πεδίου και μιλούμε για μια μακροπρόθεσμη λύση για να επιβάση των αποτελεσματικότητα στον ΚΟΑ. Η απάντηση για μας βρίσκεται στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομίας κλίμακος για τους παραγωγούς. Και προκειμένου να λειτουργήσει η εξαίρεση αυτή στην πράξη, γύρονται ερωτήσεις από τις εθνικές αρχές και από τους καλλιεργητές. Οι βασικές λοιπόν υπηρεσίες ε, της Κομισιόν, η ΓΔ Κομπ και η ΓΔ Άγκρη δηλαδή, συνεργάζονται και συντάσσουν κατευθείαν γραμμές τους τελευταίους μήνες. Αυτές οι κατευθείας γραμμές θα βοηθήσουν τους καλλιεργητές και εκείνους που θα πρέπει να εφαρμόσουν τις εξαιρέσεις αυτές, δηλαδή τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Συνεργαζόμαστε λοιπόν στενά και μαζί τους, όπως και με τα Υπουργεία και τις Γενικές Γραμματείες Γεωργίας, ώστε να απαντούμε συγκεκριμένα στα ερωτήματα αυτά. Στο τέλος του 2013 αποστήλαμε στις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού ερωτηματολόγια σχετικά με την εφαρμογή των νέων αυτών κανόνων. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία απόψεων από τις εθνικές αρχές και από τις ενώσεις των κρατών. Το οποίο δεν είναι έκπληξη γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο για τους κανόνες. Τονίζουμε όμως ότι χρειάζεται μια ενεργοντζένη προσέγγιση και έτσι η στόχευσή μας είναι πρακτικά ζητήματα, ζητήματα που έχουν σημασία στην πράξη για να εξασφαλιστεί μια ασφάλεια δικαίου και μια ενεργοσμανή προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ζήτησε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Οι νέοι κανόνες λένε ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει εξαίρεση εφόσον δημιουργεί συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα. Χρειάζεται λοιπόν να καταμετρήσουμε το κόστος και τον όγκο. Τι όγκος καλύπτεται από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικός όγκος. Αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης, γνωρίζουμε ότι πολλές ενώσεις πολλούν προϊόντα των μελών τους, αλλά και άλλα προϊόντα. Και αυτό προκειμένου να ανταποκριθούν σημαντικές υποχρεώσεις απέναντι σε μεγαλύτερους αγοραστές αυτό στι αεροτρές καλλιέργειε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι κατευθυντέ γραμμέ, λοιπόν καλύπτουν και το θέμα αυτό των προϊόντων που δεν είναι μέλη. Επίση, έχουμε το θέμα τη εξωτερική ανάθεση. Γιατί πολύ συχνά ανατίθεται εξωτερικά η μεταφορά για παράδειγμα. Αυτό ισχύει και του τρει τομεί. Και εκεί έχουμε λοιπόν καθοδήγηση για το πώ μπορεί να λαμβάνει την υπόψη αυτό ειδικά με την αποτελεσματικότητα που πρέπει να έχουμε στο τέλο. Αυτά είναι κάποια λίγα παραδείγματα θα πρέπει αυτά να ισχύουν για τους καλλιεργητές, τις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Και να αναφέρω και κάποια σημαντικά στοιχεία στο χρονοδιάγραμμα. Προβλέπονται τα εξή αυτή τη στιγμή. Έχουμε συνάντηση της Κομισιόν με τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και τα Υπουργεία Γεωργίας στις 16 Οκτωβρίου. Μετά η Κομισιόν θα πάει σε μια δημόσια διαβούλευση από την αρχή του 2015. Κατά τη διάρκεια του 2015 θα υπάρξει δεύτερη επίσημη δημόσια διαβούλευση ώστε να υιοθετηθούν οι κατευθυντικές γραμμές πριν από το τέλος του 2015. Ελπίζω αυτή η σύντομη παρουσίαση να σας έχει δώσει μια συνολική εικόνα, μια πρώτη εικόνα εν πάση περιπτώσει, της δουλειάς ε, που έχουμε θέσει επιτέπητος και περιμένω, είμαι στη διάθεσή σας για να συνεργαστώ μαζί σας ε, επί του θέματος αυτού να πάω τώρα επιτρέψτε μου στο άλλο θέμα. First of all, uh, we have to ask... Καταρχήν, uh, γιατί κάνουμε μια μελέτη για τον τομέα της λιανικής πώλησης. Η Επιτροπή έχει λάβει σχόλια από την uh, Αλυσίδα Τροφίμων και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συγκέντρωση στον τομέα και οι καταγγελίες είναι ότι οι, ιδίως ε, οι μεγάλοι λιανοπολιτές ε, ε, επιβάλλουν πολύ βαρύ όρου στου παραγωγού, και αυτό μειώνει τη δυνατότητα επιλογή και την καινοτομία ε, σε προϊόντα για, του για τους καταναλωτές. Το Δεκέμβριο του 2012 λοιπόν η Επιτροπή ξεκίνησε μία ε, σφαιρική μελέτη στον τομέα λιανικής πώληση για να δει τι έχει γίνει την τελευταία δεκαετία για του ε, παραγω... για στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θέλαμε να δούμε ποιοι ε, παράγοντες ε, καθοδηγούσαν την επιλογή και την καινοτομία. Αυτή η μελέτη είναι εντελώ νέα μελέτη. Ποτέ δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο σε τέτοιο επίπεδο και, σε, και τόσο εμπεριστατωμένη μελέτη. Καλύπτει ποικίλε περιστάσει σε τοπικό επίπεδο με διαφορετικά είδη ε, εμπορικών καταστημάτων, διαφορετικέ περιφέρειες, διαφορετική συγκέντρωση προμηθευτών και λιανοπολιτών. Περιλαμβάνει τελικά όλους τους Ευρωπαίους ε, λιανοπολιτές, όλο το λιανικό εμπόριο. Και τονίζω ότι αυτό το οποίο ε, συζητάμε σήμερα δεν καλύπτει ε, την, το σύγχρονο, τη σύγχρονη συγκέντρωση στο λιανεμπόριο. Το 1 τρίτο των κρατών μελών που έχουν υψηλή συγκέντρωση λιανικού εμπορίου δεν είχαν επαρκή δεδομένα. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη όπου υπήρχαν δεδομένα, μπορούσαμε να έχουμε κάποια εύλογη βεβαιότητα για τα στοιχεία. Θα σας απαριθμίσω λοιπόν τα κράτη-μέλη που δεν καλύπτονται από τη μελέτη. Οι σκανδιναβικές χώρες, χώρες της Βαλτικής, Κύπρος, Αυστρία, Λουξεμβούργο και Ιρλανδία. Δεν καλύπτονται αυτές οι χώρες λοιπόν από το δείγμα της μελέτης. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ότι η επιλογή αυξάνεται την τελευταία δεκαετία, αλλά μετά την κρίση επιβραδύνθηκε. Αυξήθηκε ο αριθμός των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και ο αριθμός προμηθευτών. Η καινοτομία αυξανόταν μέχρι το 2008, αλλά μετά άρχισε να μειώνεται. Η εξήγηση είναι η επιδίνωση του οικονομικού κλίματος από το 2008 και μετά. Επίσης, σημειώνουμε ότι σε τοπικό επίπεδο η δυναμική του ανταγωνισμού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί το άνοιγμα νέων καταστημάτων σχετίζεται με μεγαλύτερη καινοτομία και μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής. Πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Σε αυτή τη γραφική παράσταση βλέπετε διάφορους καταναλωτικούς τομείς με την αύξηση των εμπορικών καταστημάτων που τα έχουμε αναλύσει αναχρονική περίοδο με κίτρινο 2004-2008, με σκούρο γκρίζο 2008-2012 και μέσος όρος ε, στο ανοιχτό γκρίζο. είναι ενδιαφέρον ε, να δούμε ότι ιδίω στις αγροτικές περιοχές αυξήθηκε η δυνατότητα επιλογής για τους καταναλωτές, ιδίω στις περιοχές της Υπέθρου. Και εδώ πάλι βλέπουμε τη δυνατότητα επιλογής ε, που αυξήθηκε όσον αφορά το κατακεφαλήν εισόδημα και ως Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουμε ότι είναι πολύ θετικό ότι η μεγαλύτερη αύξηση της δυνατότητας επιλογής τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρείται σε περιοχές με χαμηλό κατακεφαλήν εισόδημα. Τώρα, τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης λιανικού εμπορίου και προμηθευτών βλέπουμε ότι σε εθνικό επίπεδο, στα κράτη-μέλη, το συνολικό ε, επίπεδο συγκέντρωσης λιανικού εμπορίου αυξήθηκε. Και, και στα σύγχρονα καταστήματα και στα παραδοσιακά καταστήματα αυξήθηκε η συγκέντρωση και στα εκπτωτικά καταστήματα που χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Στις επόμενες δύο διαφάνειες που δεν θα μπορείτε να τις δείτε γιατί είναι πολύ μικρά τα γράμματα, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, βλέπουμε όσον αφορά το τυρί, τη σχετική κατανάλωση και τη σχετική συγκέντρωση. Βλέπουμε ότι συχνά είναι προς όφελος του λιανικού εμπορίου η κατανάλωση τυριού. Βλέπουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο. Γι' αυτό η γκρίζα, το γκρίζο σχέδιο είναι πάνω από την οριζόντια γραμμή. Μόνο στην Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία βλέπουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση λιανικού εμπορίου κατά την περίοδο αυτή. Στον γαλακτοκομικό τομέα τώρα, σε αυτή τη γραφική παράσταση, παρατηρούμε ότι όταν οι αγρότες οργανώνονται σε συνεταιρισμούς, η διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι των αγοραστών, έναντι του λιανικού εμπορίου δηλαδή, αυξάνεται. Και γι' αυτό βλέπουμε το γκρίζο σχήμα κάτω από την οριζόντια γραμμή. Το προφανές συμπέρασμα είναι ότι οι μεμονωμένοι αγρότες θα πρέπει να οργανώνονται σε συνεταιρισμούς ή σε κάποια μορφή οργάνωσης. Και όπως αναφέραμε στην παρουσίαση, ο στόχος μας με τη νέα δυνατότητα που δίνεται είναι να ενθαρρύνουμε τους αγρότες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποια άλλα αποτελέσματα τώρα της μελέτης μας. Η μεγαλύτερη αύξηση ε, συγκέντρωση συνδέεται με μικρότερη καινοτομία και αντιστρόφως. Δηλαδή στις αγορές όπου η επιλογή και η καινοτομία είναι ανεξάρτητη από την διείσδυση της αγοράς των, του λιανικού εμπορίου δεν υπάρχει μεγάλη επίπτωση τουλάχιστον μέχρι να φτάσει ένα επίπεδο προϊόντος 50%. Από το 50% και πάνω αρχίζει να παρατηρείται μείωση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Oui, merci, Monsieur pour... Ευχαριστώ κύριε Σίζαρ για την παρουσίαση που κάνατε αυτών των δύο και θεμάτων. Ανοίγουμε τη συζήτηση. Έχω κάποιους εγγεγραμμένους. Ο κύριος Μισελ Νότα είναι πρώτος εγγεγραμμένος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση που μας έκανε, ειδικότερα όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, τις κατευθυντήριες γραμμές δηλαδή με τα ίδια άτομα. Είχαμε κάποιες δύσκολες συζητήσεις κατά τη σύνταξη του κειμένου για την ΚΟΑ. Ε, χαίρομαι που η ανάλυση που έγινε δείχνει ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές πρακτικές μεταξύ κρατών. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να οριοθετήσουμε, να σταματήσουμε, διότι αυτό που επιτρέπεται για τον ανταγωνισμό σε μια χώρα απαγορεύεται στη διπλανή χώρα, οδηγώντας έτσι σε, μια, σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η εργασία για τις κατευθυντήριες γραμμές είναι περίπλοκη. Ε, δίνεται μια προθεσμία που μοιάζει μεγάλη αλλά θέλουμε πραγματικά να θέσουμε στη διάθεση των αρχών ανταγωνισμού των εθνικών ένα ε, έγγραφο δράσης, ένα πλαίσιο δράσης το οποίο είναι το ίδιο για όλους. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να να καταστρέψουμε αυτόν τον ανταγωνισμό, να σκοτώσουμε αν μπορώ να το πω έτσι ε, αυτόν τον ανταγωνισμό που οδηγεί στην καταστροφή ας πούμε φρούτων που προέρχονται από μια χώρα διότι κάτι θεωρούν ότι δεν τους αρέσει. Λοιπόν, στο, όσον αφορά αυτό το πρώτο μέρος και την έκθεση που έχουμε με, ε, μελετήσει. Έχω μία ερώτηση όσον αφορά τη... τα προϊόντα ε, των διαφόρων σούπερ μάρκετ. ή διασυντικέτας δηλαδή. Είπατε ότι αυτά δεν οδηγούν σε μια αύξηση της κατανάλωσης. Είπατε ότι καμιά φορά μειώνουν τις τιμές των μεγάλων ε, ε, παραγωγών. Αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι αρνητική ειδικά αυτά τα ίδια ετικέτας προϊόντας ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οδηγούν και ε, στο σταμάτημα των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Κυρία Σαρά τώρα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτή η συζήτηση Ε, σε σχέση με τους κανόνες ανταγωνισμού είναι πάρα πολύ σημαντική για τους παραγωγούς, γυναίκες και άνδρες πρέπει να πω. Ε, εδώ και πολλά χρόνια εμείς οι εργαζόμενοι ήμασταν κάτω από πίεση στις διαπραγματεύσεις ε, και οι γεωργοί δεν μπόρεσαν λόγω των κανόνων ανταγωνισμού να διαπραγματευθούν ε, όρους ε, απασχόλησης. Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε για τους γεωργούς, άνδρες και γυναίκες, τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν τιμές που να καλύπτουν το κόστος εργασίας και παραγωγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, ο κύριος Νίκολσον. Ε, με συγχωρείτε, δεν, ε, τώρα σας άκουσα. Ε, ακολουθώ τον κύριο Ντόντον, διότι πιστεύω ότι έχει τη σωστή γραμμή εδώ. Δηλαδή, είναι μια καλή, ένα καλό σημείο εκκίνηση αυτό, αλλά η ίδια ετικέτα είναι πολύ σημαντική για τα σούπερ μάρκετ και έρχονται στον επεξεργαστή, τον μεταποιητή και του λένε είτε θα το κάνεις όπως σου λέμε ή δεν θα αγοράσουμε αυτό το οποίο παράγει. Και ορισμένες φορές οι μεταποιητέ δεν έχουν εναλλακτική λύση γιατί δεν έχουν αγορά για το προϊόν τους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε. Ε, έχουμε και ε, τους χαμένους ε, νικητές, δηλαδή έχετε ένα ελκυστικό προϊόν το οποίο σας φέρνει μέσα στο σούπερ μάρκετ σε πολύ χαμηλές τιμές και τελικά αγοράζετε και το υπόλοιπα. Δηλαδή τα σούπερ μάρκετ μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και αυτά ε, δεν είναι και πρέπει να πούμε ούτε τα κράτη, ούτε η Ευρώπη, ούτε οι περιφέρειες ε, δεν αντιστέκονται ε, μπαίνουν στην αγορά και όποιος προσπαθήσει να τους ενοχλήσει ε, απειλούν με διάφορα. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση στην οποία θα επανέλθουμε πολλές φορές και πολλές, πολύ σωστά λέτε ότι αν οι παραγωγοί δεν συνεργαστούν για να αποκτήσουν διαπραγματευτική ισχύ δεν θα τα καταφέρουν. Ε, συνεχώς όμως φαίνεται από την πλευρά της παραγωγής να υπάρχει πάντα κάποιος που θέλει να υπονομεύσει την Ένωση και να οδηγήσει σε περιορισμό των τιμών. Και βέβαια δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί αυτό. Ευχαριστώ, ο κύριος Ρόντε. Ρόντε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό στο οποίο αναφέρεται η κυρία Νίκολσον είναι ουσιαστικότατο ζήτημα γιατί θα έχετε αναγνωρίσει τι λέει η κυρία Νίκολσον και ο κύριος ε, Νταντά αλλά πρέπει νομίζω να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επέμβασή μας και στη διαδικασία μεταξύ των παραγωγών και των ε, λιανικών πολιτών. Οι παραγωγοί πρέπει να ενισχύσουν τη θέση τους. Στη Δανία έχουν συσταθεί ισχυροί συνεταιρισμοί οι οποίες έχουν καταφέρει να εξισορροπήσουν τη σχέση μεταξύ των δύο. Αλλά θα ήθελα να δω κάτι τελείως διαφορετικό. Τα θέματα ανταγωνισμού σε αυτήν την ε, ε, υλοποίηση της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι ότι δεν έχουμε θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών, διότι η υλοποίηση διαφέρει σημαντικότατα. Μεταξύ δηλαδή του τι υιοθετείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι, και τι υιοθετείται στα κρατημέλη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Πώς νομίζει ο Κομισιόν λοιπόν ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την καθυστέρηση της υλοποίησης. Γιατί ε, πρόσφατα στην Επιτροπή μας συζητήσαμε τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και νομίζω ότι είναι απολύτω σαφές ότι το όλο αυτό το στοιχείο του greening, του πρασινίσματος που λέγαμε στην ΚΑΠ, είναι ένα ένας τεράστιος διοικητικός εφιάλτης. Ένας απόλυτος εφιάλτης ε, μιας δέσμης μέτρων που είναι απόλυτα αδύνατο να δει κανείς πώς θα μπορούσε κανείς να τα υλοποιήσει. Και δεν είναι η πέτεια η Κομισιόν. Όλοι φταίνε για την ανάπτυξη αυτού του πέπλου. Πρέπει όμως να δούμε με τόσο περίπλοκους κανόνες ποιος μπορεί να τους κατανοήσει και να τους εφαρμόσει σωστά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2009 ήμουν πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Γεωργίας στην Ολλανδία και αυτά τα οποία σήμερα μας λέτε επιβεβαιώνουν την εικόνα που είχα. Η συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο ήταν πολύ σημαντική στην Ολλανδία και οι εκπρόσωποι του λιανικού εμπορίου πίεζαν ώστε να μην ισχύσουν αυτοί οι κανόνες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αλλάξει κάτι στην Ευρώπη για να μπορέσουν να είναι πραγματικότητα πλέον αυτά που συζητάμε σήμερα και να υποφεληθούν όλοι. Ευχαριστώ κύριος Βουίτεμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση που μας έκανε. Για το πρώτο τμήμα της παρουσίασης έχω μια ερώτηση. Υπάρχουν ε, νέες παρεκκλήσεις σε θέματα ανταγωνισμού και έχω ένα κάπως τεχνικό ερώτημα. Για το άρθρο 222, η χρήση αυτού του άρθρου επιτρέπει σε αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών να αποσύρουν προϊόντα από την αγορά όταν υπάρχει στρέβλωση της αγοράς. Εδώ συζητήσαμε το μποϊκοτάζ των Ρώσων. Πότε μπορεί να χρησιμοποιήσει όμως ένα κράτος αυτό το άρθρο. Πρέπει να χρησιμοποιήσει πρώτα το 219 που έχει λίγο πολύ τον ίδιο στόχο και οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Τι θα γίνει σε ένα κράτος μέλος αν κάποιες μικρές οργανώσεις παραγωγών δεν το επιθυμούν. Θέλω να πω, έχει νόημα το άρθρο 222 αν δεν είναι οργανωμένοι όλοι οι παραγωγοί σε οργανώσεις παραγωγών. Και τρίτον, κάποια κράτη-μέλη μετά το ρωσικό εμπάργο θέλουν να προσφύγουν στο άρθρο 222 για ορισμένα προϊόντα. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα εγκρίνει τα αιτήματα κάποιων κρατών μελών σχετικά με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουαζό. Κύριε Πρόεδρε, έχω δύο ερωτήσεις. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε την οργάνωση των παραγωγών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και να ρωτήσω επίσης αν το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα δίνει τη δυνατότητα να ανατρέχουν σε καλύτερες δυνατότητες προστασίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα αυτά. Καταρχάς να πω ότι Πράγματι αναφέρθηκαν κάποιοι συναδελφοί νωρίτερα. Αλλά οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το κράτος και με την περιφέρεια, να σας πω. Έχουμε λοιπόν εφαρμογή πολύ διαφοροποιημένη. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μου στην Ισπανία. Έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων αυτών ανταγωνισμού και αυτό προκαλεί στρεβλώσεις, διαφοροποιήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ε, σας ρωτώ με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή η διανομή συμπιέζει τους παραγωγούς αλλά συμπιέζει και τη δυνατότητα έρευνας και κοινοτομίας. Και εδώ είναι η ερώτησή μου πολλές επιχειρήσεις ε, παραγωγών προσπαθούν να καταβάλουν μια τέτοια προσπάθεια, αλλά περιορίζονται από την τεράστια δυνατότητα που έχουν οι μεγάλες αλυσίδες να επιβάλλουν το δικό τους εμπορικό σήμα. Οι συνεταιρισμοί προχωρούν σε προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας για νέα προϊόντα, αλλά έχουν απέναντί τους αυτήν την τεράστια δυνατότητα την απεριόριστη δυνατότητα μεγάλων αλυσίδων. Τώρα στη Ολόλαδο, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η υπερσυγκέντρωση, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε μια τεράστια ανησυχία σχετικά με τους ισολογισμούς, με την οικονομική κατάσταση των παραγωγών, με τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν παρά την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή στην Ανδαλουσία και γενικώ στην Ισπανία με τις συνεταιριστικές ενώσεις. Λοιπόν, τι ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συμφωνίες, οι διατομεακές, ή διακλαδικές συμφωνίες, πιστεύετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. κυρία Μαγκίνης. Ε, Ευχαριστώ. Νομίζω η διαφάνεια που είναι στην οθόνη είναι ενδιαφέρουσα και ε, συγκρούεται με τον εαυτό τη στη διαφάνεια αυτή, διότι στο πρώτο μέρο, ε, όπου έχουμε το τόξο μα λέει ουσιαστικά ότι η συζήτηση που είχαμε προηγουμένω για τη συγκέντρωση του λιανεμπορίου είναι άσχετη. Ε, αλλά δεν νομίζω ότι συμφωνώ λοιπόν με αυτό για την ανισορροπία και εξαρτάται εξαρτάται από το τι εννοούμε συγκέντρωση λιανεμπορίου. Αν είχαμε ένα αντίγραφο της μελέτης, ίσως θα βοηθούσε. Όσον αφορά τώρα τις ίδιες ετικέτες, και εδώ χρειαζόμαστε περισσότερες ε, μελέτες. Αλλά αν έχετε κάποιον ο οποίος πουλά αυτή τη στιγμή στο λιανικό εμπόριο, αυτό που μας λένε είναι έχουν νέες ιδέες και το πνευματικό τους κεφάλαιο το κλέβουν οι ελληνικοί έμποροι όταν βάζουν τη δικιά τους μάρκα. Βεβαίω οι αρχές ανταγωνισμού πρέπει να το διερευνήσουν, αλλά δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα, διότι ε, ε, η αρμοδιότητά σας έχει να κάνει ε, με τις χαμηλές τιμές και όχι με τη βιωσιμότητα της αλυσίδας τροποδοσίας. Ε, λέτε ότι κάνω λάθος, το βλέπω με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα σχόλιά μου, αλλά έχω άλλη εμπειρία. Μακάρι να με πείσετε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην παρουσία σας αναφερθήκατε ότι οι βαλτικές χώρες δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη σας. Κρίμα. Κρίμα διότι θα ήταν ενδιαφέρον να είχαμε και άλλες πληροφορίες για τις βαλτικές χώρες. Ίσως θα μπορούσατε να επισυνάψετε ε, μία προσθήκη στη μελέτη σας. Ο κύριος Όρλινγκ. Äh, ναι, ε, μου κάνει εντύπωση που παρουσιάζεται την κατάσταση των γαλακτοπαραγωγών ως πιο θετική τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Οι συνεταιρισμοί το ίδιο καθεστώς έχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν πολλοί συνεταιρισμοί στη Γερμανία στο γαλακτοκομικό τομέα. Ε, δεν έχουν ε, τη δυνατότητα τα μέλη του συνεταιρισμού ε, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να τα αποσύρουν για να τα δώσουν κάπου αλλού με καλύτερη τιμή. Ε, είναι λοιπόν και αυτό ένα ερώτημα. Ένας αγρότης που είναι μέλος του συνεταιρισμού έχει την δύναμη που θα ήθελε να διαπραγματεύεται για τα προϊόντα του ή πρέπει μια φορά το χρόνο να ψηφίζουν στην ετήσια συνέλευση και δεν έχουν καμία άλλη εξουσία από εκεί και πέρα. Όταν θέλουμε να προωθήσουμε τα δικαιώματα των παραγωγών, αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Υπάρχουν ε, σε πολλά κράτη-μέλη διαφορετικές απόψεις για το τι θέλουμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη θέση των αγροτών. Υπάρχει κάποια σύγκριση για τη διαφορετική εξουσία διαπραγμάτευσης των μελών συνεταιρισμών σε κάθε κράτος μέλος. Για τη Γερμανία μπορώ να πω ότι οι συνεταιρισμοί στο γαλακτοκομικό τομέα δεν βοήθησαν να πάρουν καλύτερες τιμές η παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και προτείνω να κλείσουμε εδώ τις ερωτήσεις και να δώσουμε ξανά το λόγο στον κύριο Σίζαρ για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ετέθησαν από τους βουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ομοδοποιήσω τις ερωτήσεις ή τα σχόλια τα οποία έχουν σχέση με την αποκλίνουσα εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού σε διάφορες χώρες. Πολύ αναφερθήκατε σε αυτό. Ο βασικός στόχος των κατευθυντηρίων γραμμών που επεξεργαζόμαστε σε σχέση με αυτή την παρέκκληση είναι να υπάρχει ομοιόμορφη προσέγγιση σε όλη την Ευρώπη από τις αρχές του ανταγωνισμού, ώστε να μην έχουμε αποκλίνουσες ερμηνείες ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε τέτοιες πιθανότητες. Εκτός από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, ξέρετε ότι έχουμε ένα δίκτυο αρχών ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Και προεδρεύουμε τουλάχιστον δύο με τρεις φορές το χρόνο μια υποομάδα αυτών των αρχών ανταγωνισμού για τα θέματα των τροφίμων και της γεωργίας. Προτού αρχίσουμε λοιπόν την εργασία για αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, συνεργαζόμαστε δραστήρια με τις εθνικές αρχές για να εντοπίσουμε κοινά θέματα, κοινέ προσεγγίσεις, κοινέ πολιτικές λύσεις. Τα σχόλιά σας είναι ισχυρά, τεκμηριωμένα, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερους πόρους και η ιδέα είναι να έχουμε μια ομοιόμορφη ενωσιακή προσέγγιση. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο σχόλιο της κυρίας Κίνες ότι οι αρχές ανταγωνισμοί ασχολούνται μόνο με τη τιμή και τίποτα άλλο. Το γεγονός ότι το 2012 ήδη ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη και 40 άνθρωποι και πάνω ε, εργάστηκαν για αυτή τη μελέτη σε περίοδο 18 μηνών ε, συγκεντρωθήκαμε μόνο στην επιλογή και στην καινοτομία, διότι η βιωσιμότητα και η ευημερία του καταναλωτή δεν περιλαμβάνει μόνο τη φθηνότερη τιμή, αλλά και τον τύπο της καινοτομίας που προσφέρεται. Η μελέτη είναι διαθέσιμη από την περασμένη εβδομάδα. Είναι 750 σελίδες. Είναι ό,τι πρέπει να διαβάσετε πριν κοιμηθείτε το βράδυ. Αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη δεν ασχολούμε με την τιμή. Ασχολούμεθα μόνο με την επιλογή και την καινοτομία. Και οι διαπιστώσεις είναι αυτές που ε, δημοσιεύσαμε πριν από μερικές εβδομάδες δεν ξέραμε ακόμη πώς αυτές οι διαπιστώσεις πώς θα κατέληγαν τα, αυτές οι διαπιστώσεις δεν είχαμε δηλαδή προκρίνει τα συμπεράσματα έχουμε 9 κράτη-μέλη 350 καταστήματα 100.000 ε, προϊόντα πρόκειται για μαζική συνένωση στοιχείων και κανένας μας δεν ήξερε πού θα κατέληγε. Όσον αφορά τα προϊόντα ίδιας ετικέτας, πολλοί από εσά είπατε ότι οι προμηθευτές ανησυχούν η διαπίστωσή μας είναι όταν ε, η ιδιωτική ετικέτα φτάνει σε ένα ορισμένο επίπεδο, εξαρτάται από τις κατηγορίες των προϊόντων, είναι περίπου 40 με 50%, τότε ξαφνικά ε, η καινοτομία και η επιλογή στα ράφια μειώνεται. Ε, είναι ένας συσχετισμός αυτός και η μελέτη νομίζω ότι σωστά διαπιστώνει μια, ένα τέτοιο συσχετισμό όσον αφορά τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτας. Όσον αφορά τα καρτέλ, τα, το άρθρο 222, ε, είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα. Οι αρχές ανταγωνισμού αντιμετωπίζουν τα καρτέλ κρίσης ως νόμιμο όταν υπάρχει μια ασύνηθης κρίση. Οι νόμοι πρέπει να είναι ε, εύκαμπτοι και θα ήθελα να επανέλθω ε, με μια πιο συγκεκριμένη απάντηση όταν ε, μπορέσω να συνεννοηθώ με τους ειδικούς. <coughs> Ακόμη, α, ναι, νόμιζω ότι έχω απαντήσει τα περισσότερα ερωτήματά σας για να δω τι άλλο λείπει. Όσον αφορά το πρασίνισμα, το greening, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι αρμοδιότητά μου, είναι διοικητικό βάρος σίγουρα ε, και έχουμε τους, συνάδελφου, τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη που σίγουρα μπορούν να σας απαντήσουν πιο υπεύθυνα. Όσον αφορά τα... τις τιμές γάλακτος, οι εμπειρίες μας από τον τομέα μας δείχνουν ότι αν ε, οι γεωργοί είναι εξατομικευμένοι είναι πάντα χειρότερα από όταν είναι σε μία, ένα συνεταιρισμό. Το συνεταιρισμό μπορούν να διαπραγματευτούν με μία φωνή. Τώρα, το κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, αυτό είναι σχετικό ζήτημα. Από άλλες πηγές διαπιστώσαμε ότι ένας προς ένα, ένας εξατομικευμένος γεωργός έχει λιγότερη δύναμη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι συνεταιρισμοί είναι πολύ διαφορετικοί από χώρα σε χώρα. Να, λοιπόν, και ένας άλλος τομέας που θα πρέπει να εξετάσουμε για να δούμε πιο αποτελεσματικές ε, πιο αποτελεσματική είναι συνεταιρισμή. αλλά αυτό δεν είναι θέμα του ανταγωνισμού, πρέπει να ομολογήσω. Αν έχουμε χρόνο, ε, θυμίστε μου αν ξέχασα κάτι, τις βαλτικές, α ναι, τις βαλτικές χώρες και εγώ και οι συνάδελφοι θα θέλαμε πάρα πολύ να εξετάσουμε τα εννέα κράτη-μέλη όπου έχουμε την υψηλή συγκέντρωση του λιανικού εμπορίου. Περιλαμβάνονται οι βαλτικές χώρες εκεί. Και οι κάτω χώρες περιλαμβάνονται. Δυστυχώς, τα στοιχεία, η ποιότητα των στοιχείων δεν ήταν κατάλληλη, είναι υπερβολικά αρθρισμένα και θα στη μελέτη μας ότι έχουμε πολλές πληροφορίες σε σχέση με τον τοπικό ανταγωνισμό, τι γίνεται όταν υπάρχει μεγάλη ανεργία, πώς επηρεάζονται οι επιλογές. Έχουμε πολλές πληροφορίες, αλλά δυστυχώς δεν ήμασταν σίγουροι για την ποιότητα για αυτές τις εννέα χώρες που περιλαμβάνουν και τις βαλτικές, διότι τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα. Τώρα, διερευνούμε κάποιες σκέψεις πώς θα μπορέσουμε να βρούμε τα στοιχεία. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Σε αυτές τις χώρες, αν πάση περιπτώσει για να καταλήξω, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Η κυρία Αγγιλέρα θα ήθελα να συμπληρώσει, νομίζω, την προηγούμενη παρέμβαση της. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, θα ήθελα να μου απαντήσει η Κομισιόν στην ερώτηση που έθεσα. Γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντική. Οι διακλαδικές ε, οργανώσεις και ενώσεις που έχουν προχωρήσει πολύ τουλάχιστον στη δική μου τη χώρα όπου συμμετέχουν ενώσεις παραγωγών εκπρόσωποι διαφόρων φορέων της αλυσίδας της θέσης εν εμπορία και της γεωργικής παραγωγής. Bueno. Κάτι γίνεται λέει η ομιλήτρια. Κάτι γίνεται. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Προτείνω, λέει ο Πρόεδρος, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Λοιπόν, ναι, ε, ε, κλείνω σύντομα. Για τις διακλαδικές αυτές οργανώσεις, λοιπόν, που σας έλεγα ότι ε, συμμετέχουν παραγωγή, διανομής κτλ. Φτάνουν σε συμφωνίες που είναι αδύνατο να εφαρμοστούν. Τι γνώμη έχουν οι αρχέ ανταγωνισμού σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαραματίσουν αυτοί οι φορεί. Και νομίζω ότι στη μελέτη σα αναφερθήκατε στο, αναφερθήκατε στο ελαιόλαδο. Προχωρήσαμε στην Ισπανία στην ενσωμάτωση, αλλά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κυρίαρχη θέση των μεγάλων διανομέων. Δεν ξέρω δηλαδή αν λάβατε υπαρκώς υπόψη στο ελαιόλαδο υπό την έννοια αυτή στη μελέτη σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Αγγιλέρα. Μήπως ε, ο, ο κύριος Σίζερ θα μπορούσαμε να έχουμε μία σύντομη απάντηση από πλευρά σας. Ναι, πρόεδρε. Σχετικά με τους μεγάλες κλίμακας λιανοπολιτές που ίσως να συμπιέζουν τον ανταγωνισμό και το εύρος επιλογής. Δυστυχώς η μελέτη δείχνει ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Η καινοτομία και η δυνατότητα επιλογής σε μέτρια συγκέντρωση κράτη-μέλη που συμπεριλαμβάνει την Ισπανία η επιλογή λοιπόν και η καινοτομία που καταλήγει στο ράφι για τους κατάλληλτες έχει αυξηθεί. Έχει ελαφρώς μειωθεί η καινοτομία λόγω της οικονομικής κρίσης από το 2008 και εκεί βλέπουμε το σχετισμό με τη γενικότερη οικονομική δυσκολία για τις ε, διεπαγγελματικές αυτές ε, οργανώσεις και φορείς για το πώς δρούν στην Ισπανία να σας πω ειλικρινώς ότι δεν έχω κάποια συγκεκριμένη άποψη γιατί η δική μας προσέγγιση προς τη μελέτη αυτή ήταν τι διατίθεται στα ράφια των καταστημάτων τι είδους καινοτομία φτάνει στον τελικό καταναλωτή στην περίοδο της μελέτης. Οπότε ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να κοιτάξω λίγο πιο προσεκτικά το ρόλο των ε, διεπαγγελματικών αυτών οργανώσεων στην συμφωνία και διμερώς βεβαίως ευχαρίστω είμαι στη διάθεσή σας. Λέει ο κύριος Σίζαρ. Ευχαριστούμε κύριε Σίζαρ, λέει ο πρόεδρος. Ας κλείσουμε λοιπόν τώρα και σε αυτό το σημείο και να πάμε στην τρίτη παρουσίαση για τα νέα τρόφιμα. Είναι μια γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Ο κύριος Νίκολσον εκεί είχε δουλέψει επ' αυτής της ε, γνωμοδοτήσεως. Και είχαμε την έκθεση αυτή από πλευρά τη κυρία Σάβου και θα θυμάστε από τη συνάντηση της 23 η Σεπτεμβρίου ότι η ψήφος προβλέπεται για τις 24 Νοεμβρίου επομένως αυτή η έκθεση χρειάστηκε να υποβληθεί σύντομα από την κυρία Σάβου η οποία συγγνώμη που δεν ήταν δυνατόν να παραστεί εδώ σήμερα και είναι ο κύριος Νεμπεγκά, αν ακούσαμε καλά, που θα μας ε, παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Ο κύριος Ρεμπεγκά, λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάλφοι. Ζητώ εκ νέου συγγνώμη μέρους της κυρίας Σερμπού που δεν μπόρεσε για προσωπικούς λόγους να είναι εδώ στη συζήτηση. Ε, διαβάζω λοιπόν την ανακοίνωσή της. Το σχέδιο γνωμοδότησης που παρουσιάζεται σήμερα έχει 30 τροπολογίες. Υπογραμμίζω ότι εγώ είχα μόνο λίγες ημέρες προκειμένου να προχωρήσω στο κείμενο αυτό και πρόκειται να υποβάλω και εγώ περαιτέρω ε, τροπολογίες για τα νανοηλικά, τα νέα τρόφιμα και την εξοδότηση παραδοσιακών προϊόντων τρίτων χωρών. Τον Ιανουάριο του 2008 η Κομισιόν πρότεινε τροποποίηση των κανονισμών για τα νέα τρόφιμα, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ της Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε εκείνη τη φάση συμφιλίωσης λόγω αντιβατικών στοιχείων για την συμπερίληψη νέων τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα στο πεδίο του νέου κανονισμού και σχετικά με την ιχνηλιασιμότητα ε, των ε, προϊόντων κρέατος από ακριβώς κλωνοποιημένα ζώα. Ε, το Κοινοβούλιο ζήτησε αυτό να το εξετάσουμε σε διακριτό κανονισμό. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το άκουσε αυτό και υπέβαλε προτάσεις κανονικών, διαφορετικών κανονισμών. Ελπίζω αυτά να τα δούμε ε, την ίδια χρονική στιγμή και να μην έχουμε καθυστερήσεις για την κλωνοποίηση. Εδώ έχουμε προτάσει απλούστευση τη διαδικασία εξοδότηση νέων τροφίμων, κεντρικοποιώντα τα πάντα που θα περνούν μέσω τη Κομισιόν. Δηλαδή, όλε αυτέ οι νέε αδειοδοτήσει θα υποβάλλονται, αιτήσει άδεια, θα υποβάλλονται μόνο στην Κομισιόν. Η Κομισιόν θα ζητούσε επιστημονική γνωμοδότηση τη ΕΦΣΑ. Δυστυχώ η Κομισιόν θέλει να επικαιροποιήσει μέσω ε, εκτελεστικών πράξεων, το Κοινοβούλιο ζήτησε κατεξοδότηση πράξη. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αιματήσει το ρόλο του νομοθέτη για τα νέα τρόφιμα, όπως και για τα πρόσθετα τροφίμων και τα ένζημα. Ελπίζω κατά τις ε, διαπραγματεύσει ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ληφθεί επαρκώ υπόψη και η επικαιροποιημένο κατάλογο να γίνει με διαβούλευση του Κοινοβουλίου. Για τον ορισμό δε των νέων τροφίμων, θεωρώ ότι ο ορισμό τη Κομισιόν είναι εξαιρετικά σαφή και θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση. Όπω και πρόσθετο διοικητικό άκτο για διάφορου φορεί και για τι αρχέ. Υπάρχει ο κίνδυνο για κάποια τρόφιμα που ήδη τίθενται εν εμπορία που δεν θεωρούνται νέα τρόφιμα να θεωρηθούν πλέον νέα, με τον νέο ορισμό δηλαδή που προτείνει η Κομισιόν. Από την άλλη πιστεύω ότι θα πρέπει να εισακάγουμε συγκεκριμένες κατηγορίες ε, για τους ορισμούς των νέων τροφίμων ώστε να αποφύγουμε ε, την ε, έλλειψη ασφαλείας δικαίου για όλους φορείς. Θα υποβάλω λοιπόν μια σειρά τροπολογιών που θα επανεισαγάγουν τις κατηγορίες αυτές των νέων τροφίμων με νέες προσθήκες και μιλούμε για νέα τρόφιμα όπου η μοριακή του σύσταση ή η τροποποιημένη μοριακή του σύσταση από θαλάσσια φύκια μικροοργανισμούς ή φυτικά ή ζωικά στοιχεία εκτός από εκείνα που μπορεί κανείς να λάβει μέσω παραδοσιακών ε, ε, διαδικασιών αναπαραγωγής και που έχουν και ιστορικό ασφαλούς χρήσεως και κατανάλωσης. Επίσης ε, προϊόντα εντόμων Σχετικά τώρα με τον ορισμό των ανοηλικών, αυτό πρέπει να είναι αντίστοιχο με τον κανονισμό 1169 ε, του 11. Σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, μέχρι ότου η Κομισιόν μέσω κατεξιότητας συμπράξεως ε, διευκρινίσει ε, την ανείχνευση των σωματιδίων και τη διαδικασία που χρησιμοποιείται. Πρέπει όμω να υπογραμμίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, επιταχύνουμε την ε, διαδικασία αυτή χωρί να παρεμποδίσουμε την ασφάλεια των τροφίμων. Και δεν πρέπει να έχουμε νέε προθεσμίε. Για τα παραδοσιακά δεν τρόφιμα από τρίτε χώρε η ΕΦΣΑ θα πρέπει να προχωρήσει με κατευθυντές γραμμές για τους φορείς εκείνους που θέλουν να θέσουν ε, εν εμπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραδοσιακά τρόφιμα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι φορεί συμμορφώνονται με τι ίδιε προποθέσει και απαιτήσει και το ιστορικό ασφαλούς ε, χρήσεως ε, όπως και για τα ανωτέρω. Επίσης είμαι υπέρ των γενικών αδειοδοτήσεων για τα νέα αυτά ε, τρόφιμα και υπέρ της απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ελπίζω να εργαστώ στενά, να συνεργαστώ με τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Oui, merci, monsieur. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ρέμπεκα. Αρχίζουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Μποβέ. Όσον αφορά αυτό το φάκελο νέα τρόφιμα, εντάξει, έχουμε την κλωνοποίηση από τη μία πλευρά και όλοι συμφωνούμε νομίζω ότι πρέπει να απαγορεύσουμε την κλωνοποίηση χωρίς καμία οριστία και δεν χρειάζεται να ανατρέψουμε την προηγούμενη μας απόφαση, αλλά όσον αφορά την άλλη πτυχή των νέων τροφίμων από την τεχνολογία θα αντιμετωπίσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Η αξιολόγηση δεν υπάρχει. Η ΕΦΣΑ, η Αρχή Ασφαλείας των Τροφίμων, αναγνωρίζει ότι δεν έχει τα επιστημονικά μέσα και δεν έχει τα επιστημονικά στοιχεία. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε να δεχόμαστε χωρίς στοιχεία αναλυτικά, θα οδηγηθούμε σε καταστροφή και σε έλλειψη εμπιστοσύνη των καταναλωτών το να δεχθούμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε για άδεια κυκλοφορία τροφίμων μετά από χειρισμούς νανοτεχνολογίας, αυτό δημιουργεί πρόβλημα ουσίας, ιδιαίτερα εφόσον η ΕΦΣΑ σήμερα για αυτόν τον φάκελο δεν έχει πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα για να ασχοληθεί. Θα έχουμε ένα πρόβλημα λοιπόν. Το, η εργασία που θα κάνει η ΕΦΣΑ πάνω σε αυτό θα πάρει ε, κονδύλια από άλλες δραστηριότητες της. Ε, υπάρχει ένα δεύτερο θέμα και ανησυχώ πολύ. Ε, τα αγρογεωργικά επηρεάζουν πάρα πολύ σήμερα τις νανοτεχνολογίες και οι πολυεθνικές και ο, της, του αγροδιατροφικού τομέα και ο πρόεδρος της ΕΦΣΑ ήταν μέλος γι' αυτό έφυγε, έλεγε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με την νανοτεχνολογία. Όμως ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να προστατεύσει τους καταναλωτές, διότι σήμερα κανένας δεν γνωρίζει ποιες μπορούν να είναι οι επιπτώσεις από αυτά τα νέα τρόφιμα. Για τους πράσινους λοιπόν, την ομάδα μας, είναι προφανές ότι θα αγωνιστούμε σαφέστατα σε αυτό το κείμενο για να απαγορεύσουμε σήμερα τις νανοτεχνολογίες στα τρόφιμα. Ευχαριστώ κύριε Μποβέ. Η κυρία Γιούζο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τον εκπρόσωπό της. Εγώ θεωρώ ότι η πρόταση αυτή είναι καλή. Δεν θα μιλήσω για τα κλωνοποιημένα, δεν είναι εντό τη προτάσεω. Α μην συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Μιλούμε για όλα αυτά που χρησιμοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία, μάλλον μετά την ημερομηνία δημοσίευση του του τελευταίου κανονισμού. Ο ορισμός είναι αμφίσιμος, πρέπει να τον αλλάξουμε. Και για μένα ο ορισμός είναι το αδύναμο σημείο της πρότασης αυτής. Επίσης, η κατάργηση των κατηγοριών του 208 του 97 μπορεί να οδηγήσει ένα τρόφιμα που δεν θεωρείται μέχρι τώρα νέο τρόφιμο να θεωρείται πλέον το οποίο δεν θα οδηγήσει ασφάλεια δικαίου, διότι οι φορεί είχαν συνηθίσει τι κατηγορίε αυτέ. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίε προ την κατεύθυνση αυτή. Και επίση για τον ορισμό του ιστορικού ασφαλείας επίσης πρέπει να το ορίσουμε για τις τρίτες χώρες. Γιατί και αυτό είναι αρκετά ασαφές και αφήσιμο. Πρέπει να εισαγάγουμε τις κατηγορίες και να, και να βελτιώσουμε τους ορισμούς. Σας ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για τα νέα τρόφιμα. Ε, τρόφιμα τα οποία θεωρείται ότι δεν παράγονται με παραδοσιακό τρόπο. Τελευταία φορά που το συζητήσαμε, ανέφερα ένα είδος κρέατος που πρέπει να πληρεί τις ίδιες προδιαγραφές όπως και άλλα προϊόντα κρέατος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι όμως το ίδιο γιατί υπάρχει η δυνατότητα να παρακαμφθούν οι κανονισμοί γιατί μπορεί κάποιος ε, να κουβαλήσει μαζί του στη βαλίτσα του ε, κρέας από κροκόδιλο, από φίδια και αυτά καταλήγουν και στην αγορά προς πώληση πολλές φορές και κανείς ε, δεν έχει ελέγξει τις συνθήκες υγιεινής σχετικά με τέτοια προϊόντα. Μην γελάτε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα αυτό. Θα μπορούσε ε, νεκρές μαϊμούδες να μεταφέρουν τον ιό έμπολα. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και ε, αυτοί που τρώνε τέτοιου είδους ε, φαγητό θυραμάτων ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς και δεν έχουμε και σκύλους που ανοιχνεύουν κρέας στις αποσκευές. Μπορεί να έχουμε κρέας, ε, συγγνώμη, σκυλιά που ανιχνεύουν ναρκωτικά στις βαλίτσες, αλλά όχι κρέας. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν που επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή ε, ε, η παράνοια όταν έχουμε ανάμιξη ε, σπόρων ε, σόγιας ε, γενετικά τροποποιημένων με μη γενετικά τροποποιημένους που θεωρώ ότι είναι έγκλημα. Oui, merci. La parole à madame. Ευχαριστώ. Κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Όπως έχω ήδη πει, και αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συνεδρία σε αυτό το θέμα, εμείς ε, θέλουμε να απαγορευτούν τα τρόφιμα που, έχουν, ε, που είναι προϊόν νανοτεχνολογίας. Χρειάζεται η απαραίτητη προφύλαξη και να μην χρησιμοποιούμε προϊόντα νανοτεχνολογίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτός από το γεγονός ότι η πρότασή σας σημαίνει και πάλι απώλεια κυριαρχίας για τα κράτη-μέλη. Φοβόμαστε ότι αυτή η διάταξη ε, για τις τρίτες χώρες θα επιτρέψει την εισαγωγή προϊόντων που θα ανταγωνιστούν με εθνικά προϊόντα και θα τα υποκαταστασίσουν. Χωρίς να μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα καθώς η ατλαντική αγορά ε, θα επιτρέψει την εισαγωγή προϊόντων που δεν ερχόντουσαν στην Ευρώπη. Ακόμη, οι πιέσει ορισμένων πολυεθνικών θα μπορούσαν να είναι ισχυρές προς την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γλέζος. Έχω τη γνώμη ότι τα νέα τρόφιμα πρέπει να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η κατηγορία από άλλες χώρες αλλά και η κατηγορία από τις χώρες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρώτη κατηγορία από άλλες χώρες πρέπει να βρούμε τρόπο και θα ήθελα απάντηση για αυτό πώς αντιμετωπίζεται ώστε τα τρόφιμα αυτά να είναι ανώθευτα εντελώς. Να είναι εντελώς γνήσια. Δεύτερον, να μην είναι κλωνοποιημένα Τρίτον, να αναφέρεται επακριβώς η γνησιότητα του χώρου παραγωγής είναι από την τάδε χώρα, όχι από άλλη, γιατί υπάρχει ε, τρόπος νόθευσης από χώρα σε χώρα και ο τρόπος παραγωγής. Εάν δηλαδή γίνεται με σκλάβους ή με πολύ χαμηλά ημερομίσθια η παραγωγή αυτών των τροφίμων με πιο ηθικό ηθική θεοντολογία θα δεχτούμε να τρώμε αυτά τα τρόφιμα εμείς οι Ευρωπαίοι. <clears throat> Για να μην σας κουράζω το ίδιο ισχύει όλα αυτά τα τέσσερα θέματα ισχύουν και για τις χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκα προηγουμένως και ξανατονίζω το μεγάλο γεγονός επειδή τα στοιχεία θα σας αναφερθούν και τα γνωρίζετε, τη Σαντορίνη τη γνωρίζετε όλοι, βγάζει τεράστιες ποσότητες μουστου, ο μουστος πηγαίνει στην Τινησία και από την Τινησία έρχεται στη Γαλλία και στη γιορτή του κρασιού του Μπορντό δεν πίνεται Μπορντό κρασί, πίνεται μουστο από τη Σαντορίνη. Αυτό μονάχα τα λέει όλα νομίζω γύρω από το θέμα της νόθευσης των τροφίμων και γι' αυτό πρέπει να επιμένουμε σε αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Ευχαριστώ. Merci à vous, Madame Paulsen. Η κυρία Πόλσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά πρέπει να συζητήσουμε στα πλαίσια αυτού του θέματος. Ένα συγκεκριμένο σημείο που πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε είναι ότι πολλές φορές θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών, των νέων υλικών και των χειρισμών που αφορούν τις πρώτες ύλες. Σε πολλές περιπτώσεις Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να συζητάμε την δημόσια υγεία, αλλά και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ντελέη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για τις προτάσεις και θα ήθελα και μια διευκρίνηση για το θέμα της αλλαγής διαδικασιών από εκτελεστικές πράξεις σε πράξεις εξουσιοδότηση. Φοβάμαι μήπως αυτό επιβαρύνει τη διαδικασία. Εμείς θα υποβάλουμε προτάσεις για να συμπληρωθούν οι ορισμοί, ιδίως για τα νέα τρόφιμα με συγκεκριμένες κατηγορίες. Πρέπει να διευκρινίσουμε τον όρο «σημαντική κατανάλωση» και επίσης θα κάνουμε κάποιες προτάσεις, ε, κάποιες τροπολογίες για το άρθρο 27 για την ε, προθεσμία απάντησης της Επιτροπής και για το άρθρο 18 θα υποβάλουμε μια τροπολογία για τις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει το άρθρο αυτό γιατί χρειάζεται διευκρίνηση της εφαρμογής του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντελέ. Η κυρία Μόη. Grazie signor Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνούμε με τα όσα προτείνει η συγκήτρια, ιδιαίτερα σχετικά με τις εκτελεστικές και κατεξιότητες συμπράξεις για την σύνθεση των καταλόγων των νέων προϊόντων, των νέων τροφίμων. Αλλά θέλουμε στο κείμενο του κανονισμού να υπάρχουν και κάποια ζητήματα που παραμένουν ασαφή και αμφίσιμα που θα προσπαθούμε με τις τροπολογίες μας να επιλύσουμε. Η έννοια παράδοση και παραδοσιακή χρήση τροφίμου όπου θα θέλαμε να υπάρχει συγκεκριμένη μνήμα στην συνήθη καθημερινή χρήση των προϊόντων αυτών. Επιπλέον θα θέλαμε διευκρινήσεις στο τι σημαίνει σύνθεση. Πολλά συστατικά που εισάγονται από τρίτες χώρες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν και αντίκτυπο υπό την κλιματική αλλαγή και επομένως αντίκτυπο επί των καταναλωτών. Ίδιο το θέμα για τα γεννητικώς τροποποιημένα που αποκλείεται από τον κανονισμό ε, παρότι δεν γίνεται ορισμή καμία παραπομπή στα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα όπου θα μπορούσαν να εισάγονται από χώρε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε με τι οποίε έχουμε συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Θα θέλαμε αυτό το κοινοβούλιο να εκφραστεί πολύ πιο ζωηρά επί των κυρώσεων πρέπει να είναι εναρμονισμένες ώστε να μην έχουμε κενά στο σύστημα και ώστε οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ στην ιστορική αγορά να μην βρίσκουν νοθευμένα προϊόντα ή μη υγιή προϊόντα. Ένα τελευταίο ζήτημα που πρέπει να δούμε είναι η δομή και το modus οπεράντη της ΕΦΣΑ που δεν είναι καθόλου σαφές είτε επιστημονικός υπό τα πορίσματά της είτε υπό την ανεξαρτησία της. Δεν ήταν κατά λάθο εξάλλου που είχαμε και μια έρευνα διότι οι διορισμοί στην Ιταλία είναι πάντοτε πολιτικής φύσεως όχι επί τη βάση της επιστημονικής ε, ειδίκευσης, αλλά πολιτικοί διορισμοί, ώστε να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για την Ιταλία και για όλη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, η κυρία Σέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήδη τοποθετήθηκα στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο... Μάλλον, ακούω πολλούς συναδέλφους να μιλούν για νανοτεχνολογίες και ότι θα έπρεπε αμέσως να λέμε όχι απέναντι σε κάτι τέτοιο. Ε, γίνεται πολλή δουλειά στις κατοχώρες γιατί με το θέμα αυτό. Εγώ το εξέτασα προσεκτικά και έχουν προκύψει κάποιες αρκετά ελπιδοφόρες λύσεις. Προτού πούμε ναι ή όχι, πρέπει να είμαστε σίγουροι γιατί μιλούμε. Γιατί μιλούμε και για μια σπάνιδα κάποιων πρώτων υλών και άλλων υλικών που θα μπορούσαν να περιπλέξουν το θέμα. Και αν η τεχνολογία μπορεί να δεν μπορούμε εμείς να την ε, χρησιμοποιήσουμε θα πάει στη ΣΥΠΑ, στη Ρωσία ή αλλού. Η κυρία Γιώσο γιουσο ηθελε κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ήθελα κάτι να προσθέσω. Απλώς ε, έγινε ένα σχόλιο για την ΕΦΣΑ και ως υπεύθυνη επαφή με την ΕΦΣΑ στο Κοινοβούλιο πρέπει να πω ότι οι επιστημονικές ε, εκθέσεις που γίνονται από την ΕΦΣΑ γίνονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες επιστημονικούς που δεν έχουν καμία σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο της. Και επιλέγονται αυτοί σύμφωνα με τις προτάσεις που υπάρχουν για τις υποψηφιότητες. Σε αυτό παρεμβαίνει η Κομισιόν και παρεμβαίνει και το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο μας. Επομένως ε, το να σχολιάζουμε για την ε, μη ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ δεν είναι τόσο έγκυρο, θεωρώ. Κύριε Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με το άρθρο 22 λοιπόν, όπου για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα εμπιστευτικά στοιχεία. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποια στοιχεία είναι εμπιστευτικά. Και θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε και να διαγράψουμε αυτό το άρθρο, γιατί τίποτα δεν μπορεί να είναι εμπιστευτικό για τα κράτη-μέλη. Όταν πρόκειται για τα νέα τρόφιμα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξέρουν τα πάντα σε σχέση με την κατανάλωση τέτοιων τροφίμων. Αυτή η διάταξη λοιπόν θα πρέπει να είναι ή πιο σαφής ή να αφαιρηθεί από το κείμενο. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νίκολσον που είναι εισηγητής επί της ουσίας για την Επιτροπή ΕΝΒΗ προτού τοποθετηθεί η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ο εισηγητής στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Πραγματικά Χάρηκα για την ανταλλαγή απόψεων σήμερα το πρωί, παρακολούθησα πολύ προσεκτικά όσα ελέγχθησαν. Υπάρχει μια κρόαση σήμερα που αρχίζει στις 12 και 4 για τα νέα τρόφιμα και ίσως κάποιους, κάποιοι από τους κοιόδης εισηγητές που δεν είναι εδώ σήμερα θα μπορούσαν να στείλουν κάποιον να παρακολουθήσει. Τα νέα τρόφιμα συνδυάζονται με την κλωνοποίηση. Συζητάμε χρόνια γι' αυτό. Τώρα τα έχουμε διαχωρίσει το πρόβλημα που αναφέρθηκε ε, και από τον Σκιώδη εισηγητή και από την Επιτροπή ΕΝΒΗ είναι ότι από, ο τελευταίος ορισμός ήταν το 1998 για τα νέα τρόφιμα. Συνεπώς, χρειαζόμαστε πραγματικά ένα νέο ορισμό. Δέχομαι τα σχόλια που έγιναν από την κυρία Πόλσον και από πολλούς άλλους και από την κυρία προς τα αριστερά μου. Ε, ήταν πολύ σημαντικό το επιχείρημά της. Ε, θα θέλαμε την άποψη της Κομισιόν πάνω σε αυτό. Ε, δεν χαμογελούσα καθόλου όταν αναφέρθηκε ο βουλευτής για το κρέας από θυράματα, φίδια κτλ. Δεν είναι καθόλου αστείο ε, όμως δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το θέμα έχει σχέση με την νανοτεχνολογία ή τα νέα τρόφιμα. Όμως είναι πολύ ανησυχητικό διότι μεταφέρεται μέσω του κρέατος, μεταφέρονται ε, ή όπως ο έμπονα. Ευχαριστώ λοιπόν για όσα ελέγχθησαν από αυτή την Επιτροπή, τα σημειώνω και είναι σημαντικό κάποια μέλη αυτές της Επιτροπής να έχουν διασύνδεση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι επηρεάζονται και οι δύο πολιτικές. Και από την άποψη των παραγωγών είναι χρήσιμη μια τέτοια διασύνδεση των Επιτροπών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόη θέλει να επανέλθει. Ναι, σε ό,τι αφορά στην ΕΦΣΑ θα ήθελα να διευκρινίσω η συνάδελφος ε, βρήκε στο ίντερνετ ένα άρθρο όπου αναφέρονται όλες οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφέροντος ε, που αφορούν στην ΕΦΣΑ, γιατί πολύ συχνά οι ομάδε εργασία που υποτίθεται ότι πρέπει να υποβάλουν επιστημονικέ εκθέσει γίνονται από το ίδιο άτομο που συνδέεται με συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Αυτά έχουν δημοσιευθεί στο ίντερνετ και σα παρακαλώ, προτού μιλήσετε, να, να ελέγχετε τι λέτε. Τώρα λοιπόν θα παρέμβει η Κομισιόν, κυρία Μπότσι, από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και μετά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρεμπέγκα για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Μπότσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εισηγητές και τον σκιώδη εισηγητή για τα σχόλιά τους και για την πολύ χρήσιμη έκθεση που υποστηρίζει την πρόταση που επικεντρώνεται στα νέα τρόφιμα. Όπως σωστά είπατε, η πρόταση θέλει να ευθυγραμμίσει την διαδικασία άδεια κυκλοφορίας των νέων τροφίμων και είναι πολύ σημαντικό νομοθέτημα για την υποστήριξη της καινοτομία της Ευρώπης ενώ εξασφαλίζει ασφάλεια τροφίμων σε υψηλό επίπεδο. Είναι σημαντικό νομοθέτημα επίσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μια και εισάγει την, ε, την έννοια της ε, γενετικής ε, αδειοδότησης που θα είναι πολύ χρήσιμη για τις μικρομεσαίες. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας βεβαιώσω ότι ο ορισμός που είναι στην πρόταση είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής και δεν είχαμε καμία πρόθεση να διευρύνουμε. Θέλαμε να αποσαφηνίσουμε το εύρος. Ε, βλέπουμε ότι είναι χρήσιμο να έχουμε κάποιες τεχνικές συζητήσεις για να εξασφαλίσουμε ε, βεβαιότητα δικαίου για όλους τους εμπορευόμενους και για τις εθνικές αρχές, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτός ο κανονισμός θα εφαρμόζεται με τον σαφέστερο τρόπο για όλους. Συνεπώς υπάρχουν κάποια περιθώρια για τεχνική αποσαφήνιση. Επίσης υπήρχαν, ε, έγιναν σχόλια για τρόφιμα από τρίτες χώρες. Αυτά που εισάγονται πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα όπως αυτά που εφαρμοζόνται ενωσιακά. Όπως πολύ σωστά όμως παρατηρήσατε, προβλέπουμε μία διαδικασία κοινοποίησης για ορισμένα τρόφιμα τρίτων χωρών, αλλά κάτω από πολύ αυστηρούς όρους αυτά τα τρόφιμα πρέπει να αποτελούν σύνηθη διατροφή για 25 χρόνια και δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα νέων επεξεργασιών δηλαδή δεν μπορούμε να περιλαμβάνουν από τρίτες χώρες κλωνοποιημένα προϊόντα. Αυτό είναι ξεχωριστό κείμενο. Λοιπόν, τα τρόφιμα από τρίτες χώρες έχουν αυστηρούς όρους και αν υπάρχουν αντιρρήσεις ασφαλείας από τα κράτη-μέλη, αυτά τα τρόφιμα δεν μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία πλουστευμένης κοινοποίηση. Θα πρέπει να προσφύγουν στην ΕΦΣΑ για μια πλήρη αξιολόγηση. Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε τρίτες χώρες να εξαγάγουν τρόφιμα που έχουν καταναλώσει για 25 χρόνια στις χώρες τους τουλάχιστον, χωρίς να κινδυνεύει το επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρώπη. Όσον αφορά τον ορισμό των τροφίμων από τρίτες χώρες, η ΕΦΣΑ ήδη επεξεργάζεται κατευθυντήριες γραμμές για να δει τι συλλογή στοιχείων πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ετούντα. Θα υπάρξει συγκεκριμένος ορισμός λοιπόν για την εφαρμογή αυτής της έννοιας. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό των νάνο υλικών, έχω ακούσει κάποια διαφορετικά σχόλια. Ε, κάποια σχόλια λένε ότι ο ορισμός πρέπει να είναι ο ίδιος όπως για τη σήμανση των τροφίμων, για την ενημέρωση των καταναλωτών. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προσδιορισμού αποσαφήνισης ενός περίπλοκου θέματος, δηλαδή να έχουμε έναν και μόνο ορισμό, ο οποίος να επικαιροποιείται και να εφαρμόζεται στον κλάδο των τροφίμων. Και έτσι έχουμε και βεβαιότητα δικαίου για τους εμπορευόμενους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και γενικότερα, οι κανόνες γενικά για τα τρόφιμα εφαρμόζονται και η αρχή της επιφυλακτικότητας εφαρμόζεται όταν εμφανίζεται ένας κίνδυνος και η ασφάλεια δεν είναι εξασφαλισμένη. Ε, έχουμε λοιπόν τον έλεγχο υγιεινής από τα κράτη-μέλη και άλλη οριζόντια νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται για τα νέα τρόφιμα. Επίσης θα ευθυγραμμίσουμε τη διαδικασία για να έχουμε πολύ αυστηρές προθεσμίες και για την Κομισιόν και για την ΕΦΣΑ. Παρατήρησα ότι ορισμένοι βουλευτές πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη να συντομευθεί η διαδικασία καθώς οι προθεσμίες αυτές είναι μέγιστες και μαζί με την ΕΦΣΑ έχουμε δεσμευτεί να υποβάλουμε αυτή την πρόταση μόλις εγκριθεί Τώρα, όσον αφορά τις πράξεις εφαρμογής, πιστεύουμε ότι τα κριτήρια τηρούνται για τις πράξεις εφαρμογής που προβλέπονται στο κείμενο και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα κράτη-μέλη έχουν μια κεντρική ευθυγραμμισμένη διαδικασία χωρίς να χάνουν κυριαρχία διότι εξακολουθούν να είναι ενημερωμένα για όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, το περιεχόμενο των αιτήσεων, τα εμπιστευτικά στοιχεία και όταν νέα τρόφιμα εγκρίνονται με επίπεδο ασφάλειας, αυτό δεν υπονομεύει το δικαίωμα επιλογής των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λοιπόν, γενικά θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγη, τους εισηγητές για τη θαυμάσια εργασία που πραγματοποιήσανε μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα και ελπίζουμε ότι αυτό το κείμενο θα γίνει δεκτό το ταχύτερο ε, δυνατόν ώστε αυτή η ευθυγραμμισμένη διαδικασία να εφαρμοστεί και να συντείνει στην καινοτομία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Oui, merci, Madame Σας ευχαριστούμε για αυτές τις διευκρινήσεις ο κύριος ε, Ρέμπαγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της ε, κυρίας ε, Ασέρμπο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και την Κομισιόν για τις διευκρινήσεις της Κομισιόν. Η κυρία Ασέρμπου θα συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή. Θα διαβιβάσω το μήνυμα και σας βεβαιώ ότι είναι ανοιχτή για καλή συνεργασία με όλους εσάς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Προτείνω τώρα, λέει ο Πρόεδρος, προτού περάσουμε στο επόμενο θέμα, να θυμίσω την προθεσμία καταβολής, ε, υποβολής των τροπολογιών μέχρι τις 10 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Αυτή είναι η προθεσμία καθότι το σχέδιο γνωμοδότησης είναι για 5 και 6 Νοεμβρίου. Για ψήφο στην Επιτροπή ΕΝΒΗ 24 Νοεμβρίου. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 10 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να πάμε τώρα στο επόμενο ζήτημα, το σημείο 10 δηλαδή, σχετικά με τις εξελίξεις της πανέλης των χείρων της Αφρικής σε κάποιες χώρες της Βαλτικής, όπως και στην Πολωνία. Ε... Ο πρόεδρος καταφθάνει ε, ε, γιατί επιθυμούσε να παρέμβει επί του θέματος αυτού Ναι, μέχρι, μέχρι να φτάσει εδώ ο κύριος σχετικά με την εξέλιξη του, της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων λοιπόν στην ε, περιοχή της Βαλτικής και στην Πολωνία καθότι μιλούμε για μια εξαιρετικά μολυσματική νόσο με πολύ σημαντικά επίπεδα θνησιμότητος δεν έχουμε συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης αυτή τη στιγμή της νόσου. Δεν έχουμε εμβολιασμό. Από την αρχή, από το, μάλλον του έτους, δηλαδή από τον Ιανουάριο, είχαμε 39 κρούσματα αφρικανικής παλναόλης στους χείρους και 88, αν ακούσαμε καλά, μεταξύ των αγριόχειρων. Είχαμε στη Λιθουανία, Λετωνία, Πολωνία και Ιστονία όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και από ό,τι φαίνεται προέρχεται από Ρωσία μέσω Λευκορωσίας. Από τα τέλη λοιπόν Ιανουαρίου μετά την ε, επιβέωση της 24 ε, Ιανουαρίου των δύο πρώτων κρουσμάτων στη Λιθουανία η Ρωσία όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι μπλοκάρισε τις εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις εξαγωγές προς τη Ρωσία εμπαστητώσει, στα πλαίσια του εμπάργου, επί του οποίου ε, σε κάθε περίπτωση είχαμε δυνατότητα να τοποθετηθούμε. Η Ρωσία απορροφά το 25% των προϊόντων χείριου κρέατος σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα είσοδα. Και είμαστε προφανώς κατά του εμπάργου αυτού που είναι ε, μη αναλογικού και διακριτικού χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν μια επιτροπή του ΠΟΕ να συσταθεί ώστε να βρούμε μια συμφωνία στο πρόβλημα αυτό. Τώρα, προκειμένου να διαφωνήσουμε την ε, πτυχή αυτή, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βαν Γκότεν, Γενικού Διευθυντή της ε, ΣΑΝΚΟ, ώστε να γνωρίσουμε, να ενημερωθούμε καλύτερα σχετικά με την υπόθεση αυτή. Παρακαλώ, κύριε Γενική Διευθυντή της ΣΑΝΚΟ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω ότι είναι η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Είναι μία από τις τρεις ε, πιο σημαντικές ασθένειες ε, για τα προϊόντα χείρων. Έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Πάνω από 90% θνησιμότητα για τους προσβληθέντες χείρους. Η νόσος υπήρχε στην Ευρώπη, στην Ιβηρική Χερσόνησο, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 οπότε και εξαλείφθηκε. Κάποια σποραδικά κρούσματα είχαμε και στο Βέλγιο και δυστυχώς και στη Σαρδινία υπήρχαν κάποια κρούσματα που παραμένουν ενεργά. Τώρα να δούμε πώς ε, έφτασε η νόσος στην Ευρώπη. Το 2007 στη Γεωργία υπήρχαν απόβλητα τροφίμων σε ένα πλοίο από τη Μοζαμβίκη. Ζητήσαμε από τη γραμματεία να μοιράσει ένα έγγραφο με τα κρούσματα και πώς εξαπλώθηκαν από την Γεωργία βορειοδυτικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δείτε ότι η εξάπλωση έγινε μερικές φορές αργά, μερικές φορές γρήγορα, από τον νότο της Ρωσίας προς τα πάνω κρούσματα στην Ουκρανία το 2012, Λευκορωσία το 2013. Για το πώς εξηγείται αυτή η εξάπλωση, πρέπει να πούμε ότι είναι ανεξέλεγκτη η μετακίνηση των χείρων στη Ρωσία. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στη Ρωσία είναι πολύ ανεπαρκείς. Και λόγω του στρατού επίσης εξαπλώθηκε η νόσος, διότι κάποια προϊόντα χειρίου κρέατος ε, μετακινήθηκαν από τον νότο προς το βορρά της Ρωσίας μέσω του στρατού και γι' αυτό υπάρχουν και κάποια κρούσματα πολύ βόρεια στη Ρωσία. Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξηγούν την εξάπλωση της νόσου στη Ρωσία είναι και το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση ζωοτροφών με απόβλητα τροφίμων. Στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, υπάρχει τέτοια απαγόρευση γιατί αυτό οδηγεί στην εξάπλωση του ιού και έτσι ξεκίνησε ε, και η εξάπλωση του αυθόδου πυρετού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τότε που δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης στις ζωοτροφές, ε, δεν εξαπλώνονται τα κρούσματα. Επίσης, ε, το κυνήγι είναι ένα θέμα και η πολιτική που ακολουθείται στη Ρωσία για το κυνήγι ε, δεν είναι η επιθυμητή. Από το 2007 λοιπόν μέχρι το 2014 βλέπετε σε αυτά τα διαγράμματα πώς εξαπλώθηκαν τα κρούσματα από το νότο της Ρωσίας προς το βορρά της Ρωσίας. Τι κάνουμε εμείς τώρα. Ξέρουμε ότι μέσω των αγριόχειρων μπορούν ε, να μεταδοθούν τα κρούσματα στην Ευρώπη είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν εισαγωγές χείρων ή χειρίου κρέατος από την Ρωσία διότι υπάρχουν διάφορες άλλες νόσεις, ζωονόσεις στη Ρωσία. Μέσω λοιπόν νόμιμης εισαγωγής κρέατος ή ζών των ζώων από τη Ρωσία αποκλείεται να μεταδόθηκε. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς για να προετοιμαστούμε. Υπάρχει μια οδηγία που θεσπίζει τους κανόνες για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια οδηγία του 2002. Μετά το 2010 ζητήσαμε μια γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ για τους κινδύνους που σχετίζονται με την εξάπλωση στη Ρωσία και από το 2013 όταν ο κίνδυνος ήρθε πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λάβαμε κάποια προληπτικά μέτρα. Καταρχήν φορτηγά που έρχονται από τη Ρωσία πρέπει να αποστηρώνονται πριν ξαναμπούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να απολυμένονται. Παρακολουθούμε τον πληθυσμό των αγριοχείρων στην Πολωνία και στις βαλτικές χώρες με οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν πέρυσι. Επίσης, Καλύψαμε το κόστος ε, εκστρατείας ενημέρωσης στα σύνορα και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο συζητήθηκε προηγουμένως στη συζήτηση για τα νέα τρόφιμα. Όσον αφορά το κρέας θυραμάτων από αφρικανικές χώρες, σαφώς δεν επιτρέπεται η εισαγωγή θυραμάτων από αφρικανικές χώρες, ούτε επιτρέπεται να μπει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέροντας κρέας ε, αυτό υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ελέγχουν στα σύνορα τις αποσκευές των επιβατών. Δεν μπορεί βέβαια να γίνεται αυτό στο 100% των εισαγωγών, αλλά θα δείτε ότι κάθε χρόνο η Επιτροπή εκδίδει μια έκθεση για τους ελέγχους στα σύνορα και το Heathrow είναι ένα αεροδρόμιο στο οποίο φαίνεται ότι έχουμε πολλές εισαγωγές ε, θυραμάτων ε, από την Αφρική. Στείλαμε και ελεγκτές στα σύνορα στις τρεις βαλτικές χώρες, ε, ούτως ώστε να υπάρχουν, σχέδια αντιμετώπισης των προβλημάτων και σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να επέμβουν. Βασικό στοιχείο στην πολιτική πρόληψη είναι οι κατευθυντήριες γραμμές ε, για τους αγριόχειρου που εκδώσαμε στις αρχές του 2014. Εκεί αναφέρονται σαφώς τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη έναντι ε, των ε, αγρίων ζώων τα οποία μπορούν να μεταφέρουν ε, ζώων όσους και ο έλεγχος των αγρίων ζώων πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται για να περιορίζουμε την εξάπλωση των κρουσμάτων. Ε, οι πληροφορίες ε, που λαμβάνουμε από τη Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία πρέπει να πούμε ότι δεν είναι οι πλέον πλήρε και αξιόπιστες, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι πληροφορίε παίρνουμε από τη Ρωσία δείχνουν ότι υπάρχει κυνήγι αγριοχείρων, αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να απαγορεύεται. Ο καλύτερος τρόπος για την εξάπλωση της νόσου είναι ε, το να ε, γίνεται κυνήγι αγριοχείρων, πράγμα το οποίο γίνεται στη Ρωσία και Λευκορωσία. Όταν ε, προσπαθούμε να το κάνουμε πυροβολώντας ε, τα, ε, τους αγριόχειρους ε, δεν είναι αποτελεσματικό. Πρέπει τη διαχείρισή τους να την κάνουμε με πιο σωστό τρόπο. Είτε στο δάσος είτε σε άλλες περιοχές. Αυτή είναι η γνώμη των εμπειρογνωμόνων διεθνώς. Πέρυσι, μεταξύ Ρωσίας, Λευκορωσίας και Λιθουανίας, προσπάθησαν οι αρχές της Λευκορωσίας ε, να σκοτώσουν αγριοχείρους πυροβολώντας τους και γι' αυτό είχαμε κρούσματα στη Λιθουανία και στην Πολωνία και θα δείτε ότι πολύ κοντά στα σύνορα ήταν τα κρούσματα αυτά ε, και αυτό δείχνει ότι προσπάθησαν να διαφύγουν οι αγριόχειροι από τους πυροβολισμούς από την άλλη μεριά των συνόρων και έτσι πέρασαν και εμφανίστηκαν τα κρούσματα στη Λιθουανία. 24 Ιανουαρίου ήταν το πρώτο κρούσμα στη Λιθουανία και τώρα στον άλλο χάρτη που σας έχουμε μοιράσει με το μπλε, κόκκινο και ροζ χρώμα στις διάφορες περιοχές του χάρτη 27 Ιανουαρίου είχαμε το πρώτο κρούσμα στην Λιθουανία εφαρμόσαμε άμεσα τα προληπτικά μέτρα βάσει της οδηγίας του 2002 δημιουργήσαμε ζώνες αποφυγής της εξάπλωσης της νόσου είτε μέσω ζώντων ζώων είτε μέσω κρέατος την ημέρα μετά το πρώτο κρούσμα αγριοχείρων στη Λιθουανία Οι Ρώσοι, όπως είπε ο πρόεδρος νωρίτερα, εφάρμοσαν καθολική απαγόρευση όλων των εξαγωγών χείρων και χειρίου κρέατος από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια μας εξέπληξε ως κίνηση των Ρώσων και όπως είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, πρόκειται για συναλλαγές αξίας 1,4 έως 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως και πλήττονται ιδίως η Γερμανία, η Πολωνία, καθώς και η Γαλλία και η Ισπανία που είναι, που είναι εξαγωγής χειρίου κρέατος. Στην Πολωνία πρώτο κρούσμα διαπιστώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε είχαμε κάνει πολλές διμερείς συζητήσεις με τους Ρώσους ομολόγους και σε επίπεδο επιτρόπου που ο επίτροπος πήγε στη Ρωσία προσπαθώντας να πείσει τους ομολόγους του να άρουν την απαγόρευση εξαγωγής χειρίου κρέατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα, σε επίπεδο κτηνιατρικών υπηρεσιών, τι κάναμε. Έχουμε ένα κατάλογο εμπειρογνωμόνων που είναι διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο και αυτούς τους εμπειρογνώμονες τους ειδικευμένου στην Αφρικανική Πανόλη των Χείρων και στους Αγριόχειρους, τους στείλαμε κατευθείαν στη Λιθουανία και στην Πολωνία για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν και να υποδείξουν τον καλύτερο τρόπο για την εξάλληψη της Αφρικανικής Πανόλης ε, των Χείρων και Αγριοχείρων. Ήταν μια κτηνιατρική μονάδα άμεσης επέμβασης που επενέβησαν στη Λιθουανία, Πολωνία και αργότερα και στην Λετωνία και Εστονία. Η διαχείριση των αγριοχείρων είναι ο πιο σωστός τρόπος, όπως σας είπα, για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου. Σε πολιτικό επίπεδο, ομολογώ ότι είναι πολύ δύσκολο να πει ένας υπουργός ότι, δεν, ότι θα σταματήσουν να πυροβολούν τους αγριοχείρους. Γιατί οι υπουργοί θα πρέπει να πούν κάτι πρέπει να κάνουμε, άρα τους σκοτώσουμε πυροβολώντας τους. Και ήταν πολύ δύσκολο να πείσουμε εμείς τα κράτη αυτά ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα θα ήταν να μην πυροβολούμε τους αγριόχειρους, να τους αφήσουμε να πεθάνουν από μόνοι τους. είναι ο πιο σωστός τρόπος αντιμετώπισης των κρουσμάτων. Κάναμε και πολλές συναντήσεις με την Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων που μας υποστήριξε στα επιχειρήματά μας και τα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης βοήθησαν τα κράτη-μέλη στα οποία υπήρχαν κρούσματα για να κάνουν τις διαγνώσεις των κρουσμάτων. Έκτοτε συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε μέτρα επίγουσας ανάγκης και εποπτείας με οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέτος μέχρι τώρα έχουμε προϋπολογισμό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα κράτη-μέλη που επλήγησαν, όχι μόνο για την επιτήρηση, αλλά και για την σφαγή των ε, χείρων, ε, πράγμα που πρέπει να γίνει εγκαίρος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις ε, μικροκτηνοτροφίας, μικροεκτροφέων χείρων μεταδίδονται τα κρούσματα και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα εξαπλωθούν τα, κρούσματα από τους αγριόχειρους ε, στους χείρους. Η Εστονία ήταν το τελευταίο κράτος μέλος στο οποίο υπήρξε ένα κρούσμα. 8 Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε ένα κρούσμα σε αγριόχειρο. Πάλι κοντά στα ρωσικά σύνορα, σε μια περιοχή όπου σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες που κατέφτασαν επιτόπου, πάνω από 9% του πληθυσμού είναι ε, ε, Ρώσοι και ε, αυτή ε, ε, η Ρωσικοί καταγωγοί Εστονοί κάνουν πολύ συχνά ταξίδια προς τη Ρωσία και αυτό εξηγεί την εξάπλωση με κρούσμα στην Εστονία. Στο χάρτη που σας μοίρασα με κόκκινο χρώμα βλέπετε περιοχές όπου είχαμε κρούσματα αγριοχείρων όπως επίσης και κρούσματα σε μικροεκτροφής αγριοχείρων. Με ροζ χρώμα είναι περιοχές όπου είχαμε σποραδικά κρούσματα αγριοχείρων. Και γύρω-γύρω υπάρχουν οι περιοχές με μπλε που είναι ένα είδος ζώνης προστασίας για να αποφεύγουμε την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Υπάρχουν περιορισμοί μετακίνησης από τη μία περιοχή στην άλλη, σε αυτά τα τρία χρώματα, για να προστατευτεί και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πριν κλείσω την παρουσίασή μου, κύριε Πρόεδρε, να επαναλάβω ότι επαγρυπνούμε για να αποφύγουμε την εξάπλωση της νόσου έξω από αυτές τις περιοχές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε τις αρχές να ακολουθήσουν το σωστό τρόπο διαχείρισης των αγριοχείρων και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η νόσος θα παραμείνει σε αυτές τις περιοχές όπου έχουμε θέσει τους κατάλληλους περιορισμούς. Αν προκύψουν κρούσματα στην περιοχή που βλέπετε με μπλε χρώμα, θα μετακινήσουμε αυτή τη ζώνη προστασίας για να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ελεύθερη από την νόσο. Θα θυμάστε ότι η ανάλογη πολιτική χρησιμοποιούσαμε και για άλλες ζωνώσεις στο παρελθόν. Θέλουμε να κρατήσουμε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, την νόσο και να μπορεί και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει εμπορικές σχέσεις με άλλες τρίτες χώρες. Κάποιες ε, τρίτες χώρες κάνουν εισαγωγές κρέατος από την Πολωνία, από τις περιοχές που δεν έχουν πληγεί από την όσο και θέλουμε να διατηρήσουμε τέτοιες εμπορικές σχέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Βαν Χότεν. Περιμένουμε την άφηξη μάλλον έφτασε στην αίθουσα ο πρόεδρος Σικέσκι και παρακολουθεί με ενδιαφέρον και αγωνία τη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ τώρα. Η κυρία... Uh, thank you, Mr. Παλμέντε. Yeah. Ε, Mr. President, dear Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Από την αρχή του έτους έχει εξαπλωθεί η σε αυτή της αφρικανικής πανόλης ε, των χείρων στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην οικονομία και στους καλλιεργητές μας. Εάν δεν σταματήσουμε την νόσο, η οικονομική ζημιά για το σύνολο της Ευρώπης θα είναι πολύ σημαντική. Μέχρι στιγμής οι τέσσερις χώρες που έχουν κρούσματα έχουν λάβει κάποια αποτρεπτικά μέτρα για την περαιτέρω εξάπλωση και έχουν ορίσει μια ζώνη προστασίας ε, έναντι του υπολείπου του εδάφους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά λοιπόν με την απειλή εξάπλωση σε άλλες περιφερειές και περιοχές και τον αυξανόμενο κίνδυνο της εξάπλωσης αυτής, πρέπει να λάβουμε κοινά μέτρα εκρίζωσης γιατί μιλούμε για 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τρεις χώρες της Βαλτικής. Είναι μια τεράστια καταστροφή, ένας τεράστιο κίνδυνος. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να συντονίσει τα μέτρα εκρίζωσης της νόσου αυτής για να εξασφαλίσουμε επίσης 100% χρηματοδοτική στήριξη όπως προτείνει και ο κανονισμός 652 σχετικά με την, ε, τον έλεγχο, την επιτήρηση και την εκρίζωση της αρκινικής πανόλης. Χρειάζεται επίσης 100% ε, στήριξη σχετικά με αντιστάθμιση ζημιάς, σχετικά με το κόστος ανάληψης μέτρων, καταστροφή ζωοτροφών, πρόσθετων ζωοτροφής και διαφόρων ε, φαρμάκων. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάνω έκκληση προς όλους εσάς να τονιστεί αυτό το θέμα στις υπηρεσίες της ΓΔΑ Άγκρη και όποτε βρίσκεστε με εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με αυτό το 100% επίπεδο χρηματοδοτικής στήριξης για να καταπολεμήσουμε και να εκριζώσουμε την όσο αυτή σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Βουζεκόσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρώτη. Νομίζω ότι και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω απολύτως με την κυρία Καλνιέτε. Τα μέτρα που έχει λάβει η Κομισιόν είναι ανεπαρκή. Και πιστεύω ότι η Κομισιόν δεν έχει εκτιμήσει σωστά τον κίνδυνο αυτό. Είναι κίνδυνος για το σύνολο της Ευρώπης, η νόσος εξαπλώνεται ταχύτατα για να λάβει μέτρα πάρα πολύ αδύναμα έναντι του φαινομένου. Χρειάζονται μέτρα στήριξης για τα κράτη-μέλη και τους ε, καλλιεργητές. Γιατί είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα έχουμε κρούσματα και σε άλλα κράτη-μέλη, εκτός από τις υφιστάμενες αιστείες της τέσσερις χώρας. Νομίζω ότι μιλούσαμε για κάποια εκατομμύρια στις πολωνικές ζώνες ή... Δηλαδή αυτά τα επίπεδα τιμών δεν είναι τίποτα μπροστά στην πτώση των τιμών. Και θα ήθελα επίσης να υποβάλω το ερώτημα πώς ε- ήταν δυνατό να εξελιχθεί η κατάσταση με τον τρόπο που εξελίχθηκε, καθότι τα κρούσματα αυτά προήλθαν από τη Ρωσία. Τη στιγμή κατά την οποία η Ρωσία ε, μας ε, βάζει εμπάργκο. Γιατί η Κομισιόν δεν μπορεί να αντιδράσει απέναντι σε αυτήν την ε, στάση με έναν τρόπο αποφασιστικό. Και προσθέτω το εξή με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί η Κομισιόν. Γνωρίζουμε ότι επιβάλλονται διακριτικές μεταχειρήσεις ακόμη και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η συγκεκριμένη επιχείρηση μεταποίησης του κρέατος δανική χρησιμοποιεί τέτοιες πρακτικές, δηλαδή δεν αγοράζει κρέας ε, χείριο από ζώνες που υποτίθεται ότι έχουν τέτοια κρούσματα. Εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτήν την τακτική σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ουίτεμα. Yes, thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Κομισιόν. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο συνάδελφος Κτσόφσκι. Πιστεύω ότι είναι απίστευτο η Ρωσία να είναι η πηγή αυτής της νόσου και να έχει κλείσει τα σύνορά της για το κρέας το χείριο από την Ένωση που είναι ελεύθερη από αυτή την νόσο και μάλιστα 7 μήνες πριν από το καινούριο εμπάργο. Γελία όλα αυτά. ερώτηση προς την Κομισιό. Μέτρα ελέγχου και πρόληψης εφαρμόζονται για την πανόλη των χείρων όπου υπάρχει πόνοια ή επιβεβαίωση. Ποια θα είναι τώρα τα μέτρα της Κομισιόν αν τα μέτρα αυτά δεν είναι επαρκή. Δηλαδή είναι κομμάτι του κτηνιατρικού ταμείου αυτή η νόσος όσον αφορά τον εμβολιασμό. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αποκτήσουμε ένα εμβόλιο κατά της νόσου αυτής και τι θα κάνει η Κομισιόν για να επισπεύσει Την Ιατρικό Ταμείο πάλι πιστεύετε ότι είναι παρκές για να προλάβει την διασπορά αυτής της Γνώση. στην Ένωση. Έχει η Κομισιόν υπολογίσει ή εντάξει κάποια σενάρια τα οποία μπορεί να εμφανιστούν στην Ένωση. Ευχαριστώ ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που περιλάβατε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Είναι σημαντικό να συζητούμε αυτά τα θέματα και να αποφασίζουμε τι πρέπει περαιτέρω να πράξουμε. Προσωπικά ζω κάπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Λευκορωσίας που είναι στο κόκκινο κομμάτι των εδαφών και ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. τα μεγάλα αγροκτήματα ένα δανέζικο αγρόκτημα το οποίο απασχολούσε περίπου 30 άτομα έχει κλείσει τώρα λόγω της εμφάνισης αυτής της νόσου μπορούμε να δούμε ότι όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε την νόσο εξαπλώνεται η νόσος μάλλον είναι προφανές ότι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι στις βαλτικές χώρες και στην Πολωνία υποφέρουν από αυτό και ακόμη λόγω το, της απαγόρευσης της ρωσικής στις εξαγωγές ε, παρόλο που, δεν, που η Ρωσία είναι η πηγή της νόσου. Πρώτα αρχικά όμως η σύσταση ήταν να θανατωθούν όλοι οι χείροι στη, στα αγροκτήματα, αλλά καμία αποζημίωση, αυτό έχει γίνει, αλλά καμία αποζημίωση δεν έχει δοθεί. Τώρα, η επεξήγηση είναι ότι δεν έχουν αποφασιστεί ακόμη οι λεπτομέρειες, δεν έχουν συναυτεί οι σχετικές συμφωνίες κτλ. Ένα άλλο πάλι πρόβλημα είναι το μέλλον αυτού του τομέα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν, να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα περαιτέρω, να ψάξουν διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σου, ε, ε, να αναζητήσουν διαφοροποίηση ή τι έχει τέλο πάντων το μέλλον για αυτούς. Ένα από τα μέτρα που σχεδιάστηκε από τη Λουθουγεννία ήταν να δημιουργηθεί ένας φράχτης κατά μήκο των ρωσικών και λευκορωσικών ε, συνόρων. Στην αρχή η Κομισιόν συμφώνησε με αυτό το μέτρο, αυτό το μέτρο, μετά άλλαξε άποψη και τώρα κατηγορείται η Λιθουανία για την επέκταση της νόσου και την εξάπλωση. Μπορούμε ε, να καθόμαστε και να περιμένουμε όσο του είπαν όλοι ήταν χείρον φτάσει στο Βελίο να μένουμε ακίνητοι δηλαδή και να μην κάνουμε τίποτα. Το πρόβλημα είναι πραγματικά σοβαρό και χρειάζονται και σοβαρά μέτρα. Δεν μπορείτε μόνο να παραμένουμε σε συστάσεις, να μην πυροβολούμε αγριόχειρους, να μην κυνηγάμε δηλαδή αγριόχειρους. Τι σημαίνει αυτό, ότι καθόμαστε και περιμένουμε ε, ώσπου να πεθάνουν ε, από την όσο. Η κτηνιατρική υπηρεσία της Λουθουανίας έχει υποβάλει διάφορες προτάσεις στην Κομισιόν, αλλά η Κομισιόν δεν λαμβάνει κανένα μέτρο ή δεν κάνει τίποτα με αυτές τις προτάσεις. Πρέπει να γίνει σαφής ε, ποια είναι η κατάσταση. Οι αποζημιώσεις πρέπει να καταβληθούν. Ευχαριστώ. Αλτό Μασέρα. Κύριε Πρόεδρε, παρακολουθώ αυτά που λέγονται. Και βρίσκομαι στο 1987 ξαφνικά. Ήμουνα τότε πρόεδρος κάτω χώρες στον τομέα των Χίριο. Το, το 1998 είδα ήδη ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε την κατάσταση πολιτικά. Όταν βλέπω τι συμβαίνει στη Ρωσία και τις, την, τον αντίκτυπο στις εισαγωγές είναι σημαντικό αυτό αλλά έχει σχέση και με όσα έχουν συμβεί στην Ουκρανία. Οπωσδήποτε υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα, αλλά τι να κάνουμε, να υποστηρίξουμε την πρόληψη. Ε, κυρία Κενετέ, υποστηρίζω το σχόλιο σας, όμως ο εμβολιασμό και τα μέσα που αφιερώνονται είναι το σημαντικό πράγμα. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα, η Ρωσία έχει θανατώσει χείρους, ε, έχουν πάει επιτόπου άνθρωποι, ε, η μυρωδιά είναι φοβερή στα δάση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στη Γερμανία, στην Πολωνία υπάρχουν κυνηγοί και αυτοί οι αγριόχειροι θα περάσουν τα σύνορα. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Πώς θα διαχειριστούμε το κυνήγι ε, από την ώρα που ε, θανατώνονται αυτοί οι αγριόχειροι κάτω από το κυνήγι τι θα κάνουμε. Δεν θα πρέπει όλοι αυτοί οι αγριόχοι να συνεχίζουν να πηγαίνουν προς το κέντρο της Ένωσης. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Είμαι πρόεδρος της συνεδρίασης και δίνω το λόγο στον πρόεδρό μας, τον κύριο Συρκάσκη. Έχω μία ερώτηση, την οποία θέλω να απευθύνω στην Κομισιόν. Την εξής. Πώς αξιολογείτε την κατάσταση προετοιμασίας της Ευρώπης σε σχέση με τους κινδύνους, τους υψηλούς που έχουν εμφανιστεί. Σήμερα χρειαζόμαστε να θανατώσουμε παραδείγματος χάρη μερικές χιλιάδες χείρους. Ε, είμαστε προετοιμασμένοι σε αυτό για μια τέτοια ενέργεια στην Ευρώπη. Βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλο το πλαίσιο, όλες τις προετοιμασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και κατά το παρελθόν. Αλλά σήμερα, ε, εν ώψη της κατάστασης, είμαστε έτοιμοι για μια τέτοια πράξη να θανατώσουμε ένα μεγάλο αριθμό χείρων. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο τώρα. Η διαχείριση των, του άγριου πληθυσμού δεν είναι μόνο θέμα για τους ακριόχειρους. Έχουμε και άλλα ζώα. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένε χώρες περιορίζουμε τον αριθμό ε, θυραμάτων για λόγους ανθρωπιστικούς. Αυτή η υποτιθέμενη λοιπόν ευαισθησία τελικά στρέφεται κατά των άγριων ζώων των ίδιων. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε μία αρμηνία αποδεκτή κοινωνικά, η οποία όμως θα επιτρέψει να επιλύσουμε το πρόβλημα και η οποία θα συμβάλλει στην δασική στρατηγική που επεξεργαζόμαστε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Βανγκούτεν. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Καταρχάς, φαίνεται ότι να κυκλοφορεί η ιδέα ότι δεν έχει συντονίσει επαρκώς τα μέτρα αυτά η Κομισιόν. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό. Τα τελευταία 20 χρόνια Ποτέ δεν έγινε τέτοιο συντομισμός καταπολέμησης όπως σε αυτή την περίπτωση. Κάθε εβδομάδα στέλνουμε εμπειρογνώμονες στο πεδίο για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να επανέλθω στους αγριόχειρους, του οποίους αναφερθήκατε πολύ από εσάς. Γνωρίζουμε ότι τα επίπεδα θνησιμότητας είναι στο 90%. Ο καλύτερος τρόπος να ελέγξουμε τους πληθυσμούς αγριοχείρων... είναι να τους διατηρήσουμε εκεί που βρίσκονται για να μην έρθουν σε επαφή. Γιατί η νόσος, η νόσος ίδια σκοτώνει κατά πέντε φορές πιο αποτελεσματικά τους χείρους παρότι η θανάτωση. Η θανάτωση με πυροβόλα όπλα. Γιατί όταν πυροβολούμε είτε διασκορπίζονται οι πληθυσμοί οι αγριόχειροι δεν είναι ανόητα ζώα δεν είναι έχουν μη γελάτε διασκορπίζονται οι πληθυσμοί όταν υπάρχουν τέτοιες ενέργειες και πρέπει να τους διατηρούμε συμπαγής... εκεί που βρίσκονται με διαχείριση του πληθυσμού σε μερικές περιπτώσεις και με τροφή του πληθυσμού για να αποφύγουμε να φύγουν. Μερικές άλλες φορές αποφεύγοντας να τους δώσουμε τροφή. Δεν κάνουμε τα ίδια πράγματα σε δασόδη έκταση με αυτά που κάνουμε σε μια έκταση ακάλυπτη από δάσος. Δεν κάνουμε το ίδιο για να θρέψουμε τους αγριόχειρους το χειμώνα ή άλλες εποχές του έτους. Και για να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τα τη μελη Οργανώσαμε συνάντηση την επόμενη εβδομάδα στη Λιθουανία που θα εκπροσωπούνται τα τέσσερα κράτη με τους τρεις καλύτερους εμπειρογνώμονες για τους αγριόχειρους στην Ευρώπη. Ζητήσαμε τους εκπροσώπους των ε, κρατών μελών όχι μόνο από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες αλλά και από τις, ε, τις εκπροσώπους ενώσεως ε, κυνηγών, ενώσεων κυνηγών, ώστε να είναι σαφές ότι τη στρατηγική αυτή την υιοθετούν άπαντες δεν θέλω πλέον να ακούμε ότι πρέπει να τα σκοτώσουμε τα ζώα. Αυτό ξεχάστε το. Πυροβολώντας τα ζώα είναι ο καλύτερος τρόπος να εξαπλωθεί η νόσος όπως έγινε στη Ρωσία. Και εξαπλώθηκε προς το βορρά και προς τη δύση η κατάσταση. Είναι καλύτερα να μην κάνει κανείς τίποτε απολύτως παρά να πυροβολεί τους αγριόχειρους. Δεν είναι εύκολο βέβαια για τους υπουργούς να λένε δεν κάνουμε τίποτα, η εξέλιξη, η βιολογική εξέλιξη νόσου θα τακτοποιήσει το θέμα από μόνη της. Όταν θανατώνουμε τα ζώα θα πρέπει να γίνεται αυτό με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να αποφεύγουμε τη διάχυση των ε, πληθυσμών. Για παράδειγμα, όταν σκοτώνουμε τους γονείς, τα μικρά μετακινούνται σε άλλες περιοχές για να βρουν τροφή σε κάθε εποχή του χρόνου και για κάθε περιοχή συγκεκριμένη χρειάζεται διαφορετική στρατηγική. Και γι' αυτό συγκαλέσαμε αυτή τη συνάντηση τη ερχόμενη εβδομάδα για να είναι σαφέ ότι η στρατηγική αυτή την υιοθετούν όχι μόνο οι κτηνιατρικέ υπηρεσίε αλλά και όλοι οι υπόλοιποι ενεχόμενοι. Για την έλλειψη των μέτρων λοιπόν απήντησα. Δεν το δέχομαι. Επίσης, μιλήσατε για έλλειψη χρηματικής στήριξης. Πέρσι καταβάλαμε 2,5 εκατομμύρια, πριν δηλαδή από την Όσο. Φέτος μέχρι στιγμής, επί τη βάση των προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί από τα κράτη-μέλη πριν από την Όσο, 3,5 εκατομμύρια είχαμε κατανείμει στις τέσσερις χώρες. Τώρα, με την όσο εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ζητήσει από τις τέσσερις χώρες να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους, τα προγράμματα του 2014, και είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε τη χρηματοδοτική στήριξη δραματικά για να στηριχθούν τα μέτρα αυτά που υλοποιούνται. Και συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτική στήριξη για τη θανάτωση των ζώων στις ε, μικρές καλλιέργειες όπου υπάρχει επαφή των χείρων με τους αγριόχειρους όπου προβλέπουμε έως το 40% θανάτωση σε αυτές τις ε, καλλιέργειες που ονομάζουμε backyards. Αλλά αυτό προβλέπεται για την Πολωνία και η Λιθουανία. Είμαι σίγουρος ότι θα συμπεριληφθεί και για τις άλλες δύο βαλτικές χώρες. Τώρα για τη Ρωσία. Είναι σίγουρο ότι μας ήρθε η νόσος από τη Ρωσία. Και τι κάνουν, απαγορεύουν για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι απίστευτο. και δύο μήνες μετά την απαγορευσή τη ρωσική εκινήσαμε επίσημη διαδικασία επίλυσης διαφοράς στη Γενέβη. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια που στα υγειονομικά θέματα έχουμε κινήσει τέτοια διαδικασία κατά άλλης χώρας. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρά παίρνουμε το ζήτημα αυτό. Τώρα, αν υπάρχουν επαρκή σπόροι, διατηρώντας υπόψη το, το συνολικό προϋπολογισμό της Κομισιόν, ναι. Τουλάχιστον για την, τον τομέα μας, την περιοχή μας υπάρχουν επαρκή, επαρκή σπόροι και περιμένουμε και την αύξηση του προϋπολογισμού από τις κατανομές που θα γίνουν μέσω των τροποποιήσεων των, τεσσάρων, των προγραμμάτων δηλαδή των τεσσάρων χωρών. Έχουμε την αρμοδιότητα να, να λάβουμε περισσότερα μέτρα, βεβαίως. Στα κτηνιατρικά έχουμε τη δυνατότητα με τη στήριξη των κρατών μελών να υιοθετούμε οποιαδήποτε μέτρα θεωρούμε απαραίτητα για να προστατεύσουμε το υπόλοιπο του εδάφους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το κάνουμε πολύ συχνά. Θα θυμάστε τον Αυθόδη του 2001 ή τον, την κλασική πανόλη των χείρων σε Ολλανδία, Γερμανία, ε, όπου είχαμε το 98-99 που είχαμε αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκρίζωση. Εμβολιασμοί. Τρέχει έρευνα εδώ και 20 χρόνια. Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Εμβολιασμός. Ε, ξέρω ότι η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έρευνας έχει ασχοληθεί. Έχω προσωπικά την αίσθηση ότι υπάρχουν νόσοι για τις οποίες δεν θα εξευρεθεί κατάλληλο εμβολιασμό. Τώρα αν είχαμε τεράστια κρούσματα, αν είχαμε εμπαρκείς πόρους, καταρχάς ελπίζω να μην υπάρξει αυτό. Ελπίζω να έχουμε μόνο σε μικρής κλίμακος αγρικίες με λίγα ζώα Δέκα ζώα, σε αυτά τα επίπεδα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη βιοασφάλεια στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Έχουμε τα διαθέσιμα χρήματα. Επανέρχομαι στον αυθόδη του 2001, όπου η Κομισιόν κατέβαλε κάτι λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Όχι σε ένα έτος, σε τρία έτη, αλλά κατεβλήθη το ποσό αυτό. Τώρα, σχετικά με τη ζώνη προστασίας μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, ο φράχτης αυτός, το όριο αυτό, δεν το υποστηρίξαμε ποτέ σαν ιδέα θα, το, θα τον υπερβούν το βράχτη αυτό. Θα περάσουν από κάτω, από πάνω τα ζώα. Δεν μπορούμε ποτέ να εξασφαλίσουμε. Έχουμε παραδείγματα από το παρελθόν που δείχνει ότι οι κατασκευές τέτοιου είδους δεν είναι αποτελεσματικές και γι' αυτό δεν ταχθήκαμε υπέρ. Είμαστε έτοιμοι να θανατώσουμε εκατομμύρια χείρους. Όπως έλεγα νωρίτερα υπάρχουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης τα οποία εφαρμόζουν ήδη τα κράτη-μέλη. Οι ελεγκτές των IVO ήταν στο πεδίο για να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης. Οι ελεγκτές μας είπαν ότι θεωρούν το κράτη-μέλη είναι έτοιμα και εντός των εκτάκτων αυτών μέτρων υπάρχουν προβλέψεις θανάτωσης μεγάλου αριθμού χείρων. Και αν επανέλθω σε στα παραδείγματα του αυθόδους του 2001 εξ όσων θυμάμαι στο Ηνωμένο Βασίλειο θανατώθηκαν 9 εκατομμύρια κυρίως πρόβατα και στην κλασική πανόλη σε Ολλανδία και Βέλγιο 98-99 θανατώθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια χείρι σε λιγότερο από ένα έτος. Βεβαίως λοιπόν και τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα Μερικοί έχουν κινητά μέσα όπως οι βελγικές κτηνιατρικές υπηρεσίες και οι δανεινικές ε, κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κινητά μέσα, φορτηγά, οχήματα σχετικά με τη θανάτωση μεγάλου αριθμού χείρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου. Πρόεδρε, νομίζω ότι διέτρεξα όλες τις ερωτήσεις, αν όχι είμαι στη διάθεσή σας. Merci, euh. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπανκότεμ για την παρέμβασή σας και για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Ήταν σημαντικές μετά από τη συζήτηση που κάναμε. Και τώρα προτείνω να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Έγκριση των ε, συμπερασμάτων των συντονιστών. Ξέρετε ότι χθες συνεδρίασαν οι συντονιστές και έχουμε μοιράσει τα πρακτικά της συνεδρίασης, λίγο καθυστερημένα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις για τα συμπεράσματα των συντονιστών. Ο κύριος Λουαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να αντιδράσω σε σχέση με μια αθέμητη πρακτική για την ανάθεση εκθέσεων όσον αφορά τον ζωοτεχνικό τομέα. Έμαθα ότι το ΕΛΚ θα κατέβαλε ένα πόντο, ενώ εμείς είχαμε προτείνει τρεις πόντους. Δεν είναι λογικό αυτό. Θα ήθελα λοιπόν κάποια εξήγηση για την απόφαση αυτή. Oui, από την παρατήρησή σας, κύριε Λουαζό, καταλαβαίνω ότι είναι απόφαση των συντονιστών. Είναι αρμοδιότητα των συντονιστών να αποφασίζουν πώς θα κατανείμουν τις εκθέσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Εσείς φέρετε επισήμως τώρα αντίρρηση στην απόφαση των συντονιστών χθες. Είναι μια παρατήρηση απλώς, χωρίς μικρόφωνο, κύριος Λουαζό. Ωραία, σημειώνουμε την, την παρατήρησή σας λοιπόν. Πρόκειται περί παρατηρήσεως. Θα υποβάλουμε την παρατήρησή σας στους συντονιστές. Αλλά πέραν της παρατηρήσεως δεν φέρετε, δεν έχετε κάποια ένσταση προς την πρόταση των συντονιστών. Ευχαριστούμε. Άλλες παρατηρήσεις για την έκθεση των συντονιστών. Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι εγκρίνεται η πρόταση που μας υπέβαλαν οι συντονιστές. Στα διάφορα δεν έχουμε κάποιο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ πολύ και προτείνω να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστεί και του διερμηνείς ο Πρόεδρος, τον ευχαριστούν και οι διερμηνείς. Και σας υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου, 9 με 12.30 και 3 με 6.30 και στις 6 Νοεμβρίου 9 με 12.30. Θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη φορά. Γεια σας.